Αγαπητοί συνάδελφοι, καλώ ήρθατε στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ελέγχου Προϋπολογισμών. Βλέπω ότι δεν έχουν έλθει ακόμη όλοι οι συνάδελφοι. Φαντάζομαι ότι είναι λόγω της δυσκολίας μετακίνησης λόγω του χιονιού και γι' αυτό ακριβώς ε, προφανώς βρίσκομαι εγώ στην Προεδρία της συνεδρίασής μας στην αρχή της συνεδρίασης. Κύριε Οντί, δεν ακούτε γαλλικά? Α, ακούτε. Ο κύριος Τόρερ είναι κάπου ανάμεσα στην ε, πόλη του και εδώ, δεν έχει έρθει ακόμη. Εγώ θα προεδρεύσω μέχρι να έρθει. Έχουμε μια φορτωμένη ημερήσια διάταξη. Το πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη είναι η έγκριση αυτής. Υπάρχουν κάποιες προτάσεις τροποποίησης που έχουν προταθεί, το 4 για παράδειγμα, που είναι η εκλογή νέου αντιπροέδρου μετά την αναχώρηση της ε, κυρίας ε, Ιβάνοβα. Θα πάρουμε λοιπόν αντί του 4 το σημείο 10, κατόπιν αιτήματος του κυρίου Ντόιτς. 9. Συντονιστέ. Αύριο θα του κάνουμε του συντονιστέ, γιατί η κυρία Γκρέσλε, η συντονίστρια από το ΕΛΚ, δυστυχώ δεν μπορεί να είναι εδώ μαζί μα. Οπότε αύριο μετά το 14 θα κάνουμε τους συντονιστές. 15. Ειδική έκθεση θα το κάνουμε στις 20... Ε, θα το προτάξουμε σήμερα. Είστε ικανοποιημένοι με την ε, αλλαγή αυτή. Ο κύριος Γκάιερ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κοιτάξτε, στη συνεδρίαση των συντονιστών είχαμε πει ότι στην αρχή της συνεδρίασης ε, θα πρέπει να συζητήσουμε για να δούμε τι θα κάνουμε τελικά με την έκθεση Μαρινέσκου ε, για το Nuclear Decommissioning. Και ε, αν θυμάμαι καλά, η ε, Επιτροπή μας καλείται να ψηφίσει τώρα, πριν ξεκινήσει την και κατά πόσο το θέμα θα παραμείνει στην μερίσια διάταξη ή όχι. Κοιτάξτε, θα ήθελα να πούμε πρώτα, να φτάσουμε πρώτα στις ανακοινώσεις του Πρόεδρου και αργότερα να εξετάσουμε το θέμα αυτό, όπως αναφέρεται στο κόκομπι. Και θέλω να πω το εξής. Ο κύριος Τόγρα μετά από αυτή τη συνεδρίαση μας καλεί σε δεξίωση στις 6.30. Αλλά αν τελειώσουμε 6 παρατέταρτο, θα ακολουθήσει αμέσως μετά η δεξίωση. Δεν χρειάζεται να περιμένουμε μέχρι τις 6.30. Έχουμε και έναν νέο συνεργάτη, Πιότε Μπαρτότσεβιτσε Μαλίκη. Είναι δύσκολο το όνομά του, ε, τον καλωσορίζω και προσβλέπω στην αγαστή συνεργασία μαζί του. Σημείο 3. Πρακτικά της συνεδρίασης. Όποιος, ε, αν κάποιος δεν έχει αντίρρηση, εγκρίνονται τα πρακτικά. Πάμε στο σημείο υπαριθμό 5. Ειδική έκθεση, είπαμε, αναβάλλεται για αργότερα. Και πάω τώρα σε αυτό που, ανέθεσε, που ανέφερε ο κύριος Γκάια. Την προηγούμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο είχαμε συνεδρίαση των συντονιστών μετά από αίτημα των σοσιαλδημοκρατών. Και εκεί συζητήθηκε το ερώτημα κατά πόσον η έκθεση Μαρινέσκου ε, θα εξεταστεί ή όχι. Και πρέπει να πω εδώ, οι σοσιαλδημοκράτες είπαν ότι δεν πρέπει να συνεχιστεί η ψηφοφορία και οι συντονιστές της Επιτροπής πρέπει να αποφασίσουν. Δηλαδή τώρα καλούμεθα να ψηφίσουμε και θα δούμε ανάλογα ε, ή θα εξετάσουμε το θέμα ή όχι. Μήπως θέλει το ΕΛΚ να πει κάτι, όχι. Άρα ψηφίζουμε για αυτό το θέμα. Παρακαλώ να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά για να δούμε ξεκάθαρα την πλειοψηφία. Ψηφίζουμε λοιπόν για το ερώτημα κατά πόσον η έκθεση Μαρινέσκου θα πρέπει να τεθεί σε ψηφοφορία ή όχι, θα εξεταστεί ή όχι. Αν ψηφίσετε ναι, θα το εξετάσουμε το θέμα, αλλιώς θα αφαιρεθεί από την ημερήσια διάταξη. Όποιος, ε, να το πω αλλιώς, εάν η πλειοψηφία ε, υπερψηφίσει, τότε θα εξεταστεί το θέμα. Και εάν ε, Ψηφίζετε όχι, θα αφαιρεθεί το θέμα από την ημερήσια διάταξη. Ψηφίζουμε λοιπόν ηλεκτρονικά παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Ο κύριος Σκυλακάκης, ε, από ό,τι άκουσα, δεν έχει την κάρτα του, οπότε θα σας προσθέσω κύριε Σκυλακάκη. Ωραία, λοιπόν, έκλεισε η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Μήπως υπάρχει κάποιος ο οποίος ε, δεν έχει την κάρτα του. Ο κύριος Σκυλακάκης, ο κύριος Γκεμπράντη, τι ψήφισατε κύριε Σκυλακάκη, υπέρ, υπερψηφίσατε. Καλώς. Και ο κύριος Γκεμπράντη, και εσείς, και εσείς υπέρ. Δύο ναι λοιπόν πρέπει να προσθεθούν στο αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. 12-9, άρα θα ψηφίσουμε για το θέμα αυτό. Πάμε τώρα στον κατάλογο ψηφοφορίας. Ehm, eh, Συγγνώμη, Κύριε Επιτρόπε, συγγνώμη, αλλά έπρεπε να κάνουμε αυτή την ψηφοφορία πριν συνεχίσουμε. Να ψηφίσουμε, λοιπόν. Παράγραφος 1, τροπολογία 1, 2 και 3. Συμβιβαστική τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 4. Καταπίπτει 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Έξι. Ιγκεμπροπ κρέσλε. Υπέρ. Κατά. Δεν είναι σαφέ. Ηλεκτρονικός έλεγχο. Μιλάω για την Έξι Ingeborg Gressle. Αν δεν έχετε την κάρτα σας, σηκώστε τα χέρια σας. Κύριο Κυλακάκη είναι υπέρ. Κλείνει η ψηφοφορία. Εγκρίνεται 13-7. 7, 8, 9, 11, 12. Είναι συμβιβαστική 2 υπέρ. Κατά αποχέ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 10. Πρέπει να την ψηφίσουμε. Okay. Dan gaan we uh, eerst stemmen over amendement 173 van uh, de heer Balsitis. Wie stemt... Λοιπόν, ψηφίζουμε ναι το πρώτο τμήμα, υπέρ, κατά, en εγκρίνεται. Πάμε τώρα στη συμβιβαστική 3. 13, 14, 15, 16 καλύπτεται από τη συμβιβαστική 3 ε, υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 17 καταπίπτει, 18 επίσης, 19 καλφίν υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 147 παλσίτης υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 20 21 και 22 Σοντάργας υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 23 και 24 υπέρ κατά αποχές δεν είναι πολύ σαφές να ψηφίσουμε και ηλεκτρονικά μιλάω για την 23 και την 24 έναρξη ηλεκτρονικής ψηφοφορίας πέρας εγκρίνεται 28 υπέρ κατά αποχές δεν εγκρίνεται, απορρίπτεται 26 ανδρική ένε υπέρ Κα, κατά αποχές απορρίπτεται 27 δική μου υπέρ κατά απορρίπτεται Okay. You have to be faster. <laughs> Eh, eh, eh, blijkbaar hebben we een aantal amendementen gestemd die al, die al niet meer gestemd Έχουμε ψηφίσει κάποιε τροπολογίε, οι οποίε δεν έπρεπε να τι ψηφίσουμε. Τέλο πάντων. Συμβαστική 4, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 29. Την ψηφίζουμε. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 30. Συμπεριλαμβάνεται στη συμβιβαστική 3. 31 λοιπόν. Καταπίπτει. Σαράντα 46 και 46 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Να ψηφίσουμε ηλεκτρονικό 45 και 46. Ωραία, εντάξει. Ηλεκτρονικός λοιπόν ελέγχουμε 45-46. Πέρας. 10-10. Άρα οι δύο συνάδελφοι που δεν έχουν ε, την κάρτα τους, πώς ψήφισαν. Αν ψηφίζατε υπέρ θα ήταν 11-10, οπότε θα περνούσε η τροπολογία. Τέλος πάντων. 47. Καταπίπτει. Λείπει μία σελίδα από τον ε, κατάλογο ψηφοφορίας μου. Ναι, αλλά δεν ψηφίσαμε την 32-33, λέει ο συνάδελφος. Ναι, συγγνώμη, το πέρασα γιατί πήγα στην επόμενη σελίδα γιατί δεν ήταν στον κατάλογο ψηφοφορία μα. Έλειπε μία σελίδα. Ε, συγγνώμη, πήρα τον καινούριο κατάλογο τώρα που ελπίζω να είναι σωστό. Συγγνώμη, λίγη επίκεια. Την 32 λοιπόν ψηφίζουμε. Την 32. Τέλος πάντων ψηφίζουμε την 32 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Να την ψηφίσουμε και ηλεκτρονικώς. 32. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται 11-10. 34 αποσύρεται, 35 επίσης, γιατί καλύπτεται από την συμβιβαστική τρία που εγκρίθηκε. Άρα πάμε τώρα στην 37, αντρική 1, υπέρ, κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Μιλάω για την 36. Άρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία για την 36. Πέρας. 11-10. Εγκρίνεται. 37. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 38. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι απορρίβεται να ψηφίσουμε και ηλεκτρονικώς για να το ελέγξουμε. Μιλάω για την 38. Πέρας. Υπέρ. Ε, κατά. Ναι αποχές 40 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία υπερθμό 41 θα κάνουμε παλήθηση για την 40. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας αυτής. Απορρίπτεται. Τροπολογία 41. Δική μου. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Αλλά μια που θέλω να είμαι αμερόληπτος, παρακαλώ ας απελευθεύσουμε. Μια που είναι δική μου τροπολογία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας εγκρίνεται. 42 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 43 καταπίπτει. 44 δεν την έχω βρει ακόμα. Α, είναι προφορική τροπολογία 44 που καλύπτει και την 47. Η προφορική τροπολογία ψηφιπέρου. Κατά. εποχές Εγκρίνεται. 45 πρέπει να την ψηφίσουμε. Τροπολογία 45. Ζητώ τη βοήθεια της γραμματείας. Δεν, δεν είχα σκοπό να κάνω αυτή τη ψηφοφορία. Ζητάει την διαγραφή της παράγραφου 12. Συνεχίζουμε λοιπόν με τις 45 και 46. Ωραία. 45 τροπολογία. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 46. Του κυρίου Ουρουτσεφ. Α, όχι, όχι, συγγνώμη. Η 47 καλύπτεται από την προφορική τροπολογία. 48 δεν χρειάζεται να ψηφιστεί και μπορούμε έτσι να περάσουμε στην συμβαστική τροπολογία υπαρθμών 5. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Η συμβαστική τροπολογία 5. 51. Ούρουτσεφ. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές θα πρέπει να ελέγξουμε. Τροπολογία 51. Πέρα ψηφοφορίας. 11-10. Έγινε δεκτή. 52. Του κυρίου Κάλφιν. Υπέρ. Όχι, 52 και 53 καταπίπτουν. Πρέπει να είμαι προσεκτικός διότι εδώ στο έντυπο που έχω ενώπιον μου δεν είναι ξεκάθαρο τα πράγματα. 54 ψήφι Κατά αποχές δεκτή. Επαλήθευση 54. Άρχιδη ψηφοφορία. Πέρας. Ισοψηφία, άρα απορρίπτεται. 55. Ψήφι Κατά. Με αποχές. Δεκτή. Νομίζω. Ας επαληθεύσουμε όμως. Για την 56 ψηφίσουμε. Πέρας της ψηφοφορίας. Ισοψηφία. 11-11. Απορρίπτεται. 57. Υπέρ. Κατά. Νομίζω ότι έχουμε την αυτή πλειοψηφία. Ας το επαληθεύσουμε όμως. Πέρα στις εφορίες. Υπάρχει μια ομάδα από την οποία ψηφίζει ένας παραπάνω. Όχι, όχι. 12, 11 εγκρίνεται. Η επόμενη του Πάξα υπέρ κατά εποχές. Ας επαληθεύσουμε και εδώ πέρας της εφορια 12 12-11 έγινε δεκτή 61 κάλφιν υπέρ κατά αποχές η ίδια πλειοψηφία και εδώ νομίζω πως εγκρίθηκε θέλετε να επαληθεύσουμε παρακαλώ Ψηφίσατε. ψηφοριες ψηφοφορίας. 12-9 δεκτή. 62 καταπίπτει, 61 εγκρίθηκε, 64 επίσης, 65 επίσης. Περνάμε στην 66. και δεν 67 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας επαληθεύσουμε λοιπόν και εδώ. Οι διαφορε ειναι είναι πολύ μικρές. Πέρα ψηφοφορίας. 12-11. Δεκτή. Εβδομήντα δύο. και με τη 73 υπέρ κατά αποχές Η γραμματεία μου λέει πως διαγράφεται η παράγωση, άρα δεν μπορούμε να ψηφίσουμε επιτροπολογιών 72-73. Ας περάσουμε σε ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέρα ψηφοφορίας. Εγκρίνονται. 77 τροπολογία υπέρ κατά εποχές επαλήθευση έληξη ψηφοφορία δεκτή με μία ψήφο διαφορά και τώρα Μπορούμε να περάσουμε στην 84 τροπολογία ο Κάλφιν 85 και 86 ψήφι υπέρ κατά Α, θα επαληθεύσουμε. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. 12 δέκα. Πάντα με διαφορές στήθους. Δεκτή. Μητροπολιτεία 92. Κάλφιν. Με 93, 94, 95 και 96 ψήφι πέρα. Κατά. Επαλήθευση. Άρχεται την ψηφοφορία. Πέρα τη ψηφοφορία. 12-10. Η αυτή η πλειοψηφία εγκρίνεται. 98 κάλφιν υπέρ. Κατά. Αποχές. Η ε, αυτή η πλειοψηφία. Ή θέλετε να επαληθεύσουμε. Ο εισηγητής επιμένει επαλήθευση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας επαλήθευση ψηφοφορια περας 12-10. 99 υπέρ κατά καταπίπτει 100 υπέρ κατά αποχές η αυτή η πλειοψηφία με όλες τις υπόλοιπες θέλετε παλήτευση κύριε Σιγητά ή το δέχεστε το αποτέλεσμα το δέχομαι Τροπολογία 101. 102. Νομίζω ότι δεν έχουν πλέον νόημα. Περνάμε στην 103. Είναι συμβατές με την 102. Ψηφιπέρ, κατά. Αποχές. Η ίδια πλειοψηφία εγκρίνεται. 103. Τροπολογία 104 του κυρίου Ορντή. Προφορική τροπολογία ψηφιπέρ. κατά εποχές νομίζω πως ε, απορρίφθηκε αλλά θα πρέπει να το ελέγξουμε 104 προπολογία. πέρα της 814 8 8-14 απορρίπτεται έχω ένα κακοτυπωμένο έντυπο ενώπιόν μου, 107 τροπολογία, προφορική. Ψήφι υπέρ της προφορικής τροπολογίας κατά. Αποχές. Δεκτή. 105-106 είναι μας με την 104. Πρόκειται για τις αυτές τροπολογίες και καλύπτονται από την προσωπική τροπολογία του κ. Οντί. Με 104 την έχουμε εγκρίνει. σχόλια από την αίθουσα εκτός μικροφώνου. Τι έχει γίνει με την... Τι έγινε με 104. Κοιτάξτε, τροπολογία 107, τροπολογία προφορική, 105 ε, και 107 δεν χρειάζεται να ψηφιστούν. να βλέπετε μερικές φορές κάνει και λάθη και η γραμματεία και έχει δίκιο η κυρία Γιάλα, έχετε δίκιο. Κυρία Γιάλα θα ψηφίσουμε πρώτα την 105 και μετά την 106 που είναι και ταυτόσιμες ψήφι πέρου. Κατά αποχές εγκρίνεται. 107-108 προφορική τροπολογία. Πάξας Μπαχτήτης Μαξίτης ε, υπέρ. Κατά εποχές δεκτή τροπολογία 109 και 110 με το σχόλιο που έχει συμπεριληφθεί ψήφι ε, υπέρ κατά απορρίτεται. επαλήθευση εγώ είμαι κατώ σίγουρος, σε εμπεριστώσει άρχη ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορίας. 15-8 έχει απορριφθεί η τροπολογία. 176 γκάγια υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 111 αντρική 1 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 112 και 113 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 114-115 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 116, 117, 118. Αυτές τις τρεις τροπολογίες ομού υπέρ κατά αποχές ας επαληθεύσουμε 116, 117, 118 άρχιτη ψηφοφορία πέρας 12-10 το αποτέλεσμα εγκρίθηκαν 119 καταπίπτει. 174 υπέρ. Κατά. Εποχές. Εγκρίνεται. 178, 179, 180, 81, 82, 83, 184 να ψηφιστούν on block υπέρ κύριο Κυλακάκης. En bloc. Μέχρι την 183. Ψηφιστούν ο μπλοκ. Υπέρ. Κατά. αποχέ δεκτέ. 184. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Δεκτή. 120. Με αυτόν τον κατάλογο που έχω εδώ μπροστά μου τα πράγματα καθίστανται ιδιαίτερα δύσκολα. Υπέρ, κατά, εποχές, Νομίζω πως ε, εγκρίθηκε η τροπολογία. Αλλά ας επαληθεύσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα της 13 13-8 το αποτέλεσμα. Έγινε δεκτή 125 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Συνεβαστική 8 που καλύπτει 126 και έρχεται τροπολογίες ψήφι υπέρ κατά αποχές δεκτή. 185 υπέρ κατά αποχές δεκτή 128 υπέρ κατά αποχές δεκτή 129 υπέρ κατά αποχές δεκτή ε, στο θέλει επαλήθευση, όχι, δεκτή. Περνάμε στην 130 δεν χρειάζεται να ψηφιστεί διότι καλύπτεται από άλλη τροπολογία που εγκρίθηκε την 121 περνάμε στη συμβασική τροπολογία περνούμε 9 αφορά στις τροπολογίες 131-132 υπέρ κατά αποχές δεκτή 186 υπέρ κατά αποχές δεκτή Συμβαστική 10 που αφορά στις τροπολογίες 187-193 υπέρ κατά εγκρίνεται. 133 το κ. Κάλφιν υπέρ κατά αποχές δεκτή. 134 υπέρ. 134-135 είναι ταυτόσιμε Κατά εποχέ λέγεται. 136 καταπίπτει, 137-138 επίσης. 189 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 141 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 142 κάλφιν υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 143 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 144 καταπίπτει. 145 πάξας υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 146 αλφιν υπέρ κατά αποχές δεκτή 147 υπέρ κατά αποχές θα επαληθεύσουμε πέρα ψηφοφορίας 9, 14. Απορρίπτεται. 148. Μαζί με 149 υπέρ. Κατά. Αποχέ. εγκρίνεται. Πάμε λίγο παρακάτω, 190 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 53, 54. Θα ψηφιστούν χωρίς τα 153. Θάλφιν. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Τουλάχιστον έτσι κρίνω. 154 καταπίπτει. 155 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται με 191 υπέρ κατά αποχές δεκτή 156 έχει αποσυρθεί 157 επίσης ή πρέπει να τη ψηφίσουμε 157 ψήφι πέρα. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 158 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 159 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Θέλετε παλήθευση, όχι. 160 και 161. Όχι, όχι. Συγγνώμη. 160, 61, 62 καταπίπτουν. 163. Και συμβασική τροπολογία 11. 164, 165, 166 υπέρ κατά αποχές δεν ήταν σαφές το αποτέλεσμα θα ελέγξουμε ηλεκτρονικό ε, συμβαστική 11 πέρα της ψηφοφορίας 15-7 εγκρίθηκε 168 κάλφιν υπέρ και για το συμβιβασμό 11. 167 είναι κομμάτι του συμβιβασμού υπαριθμών 11. Ο συγητής, τι γνώμη έχει. Πρέπει να ψηφίσουμε και την 167, ρωτά ο πρόεδρος. Αποτελεί τμήμα του συμβιβασμού. Λοιπόν, θα ακολουθήσουμε την γνώμη του συγητή και περνάμε στην 168. Υπέρ. Κατά αποχές δεκτή 179 καταπίπτει 170 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 171 αντρική είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται πρώτη τελευταία 172 αντρική είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται και τώρα η γραμματεία με ενημερώνει σχετικά ελέγχουμε αλλά ελέγξτε τα και εσείς 88, 89 και 90 δεν ψηφίσαν αυτές τις τροπολογίες δεν ξέρω γιατί ψηφίσαμε αλλά αυτό είναι το αποτέλεσμα 89 90 Est-ce que le rapporteur peut... Μήπως ο εισηγητής μπορεί να επαληθεύσει. Δεν έχουμε ψηφίσει τις τροπολογίες 88, ε, 89 και 90. Ο εισηγητής τη φρονεί. Συγγνώμη, αλλά δεν σκόπευα να προεδρεύσω σήμερα, γι' αυτό τα πράγματα δεν ε, κυλούν ε, και πολύ ήρεμα. Τροπολογία 84 τι έγινε. Δεκτή ή απορρίφθηκε. And It's better to, to check, to check Six. Καλύτερα τώρα που ελέγχουμε. Όπως λέμε, μέλη... Κάλιο. κάλλιο γαϊδουρό δεν είναι παρά γαϊδουρό γύρευε. The, the paragraph was deleted, so there's no compromise to the paragraph. Ah. Okay. Eh, Ωραία, εντάξει. Όλα ξεκαθαρίστηκαν τώρα. Περνάμε στην τελική ψηφοφορία, ηλεκτρονικά παρακαλώ. Τελική ψηφοφορία της έκθεσης Μαρινέσκου. Άρχεται η ψηφοφορία. Ik Δεκτή 14 ψήφοι υπέρ, 8 κατά μία αποχή. Συγχαρητήρια κύριε Σιγητά. Sorry, Soms een beetje hakkelend verliep. Λυπάμαι που καθυστερήσαμε περισσότερο από όσο είχαμε υπολογίσει. Καλώ λοιπόν τον κύριο Επίτροπο να έρθει εδώ πλάι μου. Goed, collega's, we, collega's, we gaan naar punt 7 van de agenda. De gedachtenwisseling. περάσουμε λοιπόν στο σημείο 7 τη ημερησίας διατάξεω. Ανταλλαγή απόψεων με τον Επίτροπο Σεμέτα. Είναι παρόντα και δύο πρόσωπα από το ελεκτικό συνέδριο, το, των οποίων τα ονόματα μου είναι πολύ δύσκολο να προφέρω. Προτείνω να λάβει το λόγο πρώτα ο Επίτροπος ή το ελεκτικό συνέδριο. Πρώτα το ελεκτικό συνέδριο και μετά ο Επίτροπος. Ποιος θα ξεκινήσει, η κυρία Κάγιου Λάιντερ. Ευχαριστώ Πρόεδρε και που μου δίνετε την ευκαιρία να σας παρουσιάσω σήμερα επιπρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το 2011. Όπως γνωρίζετε, το κεφάλαιο 1 αποτελεί ε, το απάβγασμα των συμπερασμάτων μας, άρα δηλαδή αυτό που καλούμε εγώ να κάνω σήμερα I can continue? I promise I stay with English. Unfortunately, only Estonian, English and Finnish are. Λοιπόν, θα συνεχίσω αγγλικά. Όπως σας είπα λοιπόν, το κεφάλαιο υπαριθμών 1 είναι το απάβγασμα των ε, συμπερασμάτων μας και άρα δηλαδή εγώ αυτό που καλούμε είναι σήμερα να σας παρουσιάσω ε, στην προοπτική τους τα αποτελέσματα τα οποία έχουν παρουσιάσει διάφοροι συνάδελφοι και επίσης να σκεφτούμε από κοινού για τις ε, δυνατότητες που υπάρχουν για το μέλλον η δήλωση αξιοπιστία ε, του ε, δικαστήριου του για το 2011 περιλαμβάνει πέντε γνωμοδοτήσεις και χαίρομαι πάρα πολύ που για έκτο συναπτό έτος ε, οι λογαριασμοί γκρίθηκαν κάτι που δεν αναφέρεται συχνά. Όσον αφορά τώρα την κανονικότητα των συναλλαγών το δικαστήριο διαπίστωσε ότι δεν υπάρχει τυπικό σφάλμα και Αυτά, αυτό παρέμεινε στο ίδιο επίπεδο το τυπικό σφάλμα όπως το 2010. Επίσης, ε, οι έλεγχοι δείχνουν ότι τα σφάλματα δεν περιλαμβάνουν σε έναν ή δύο μόνο τομείς του προπολογισμού. Το δικαστήριο καταλήγει στο ότι εκτός από τις ε, ομάδες εξωτερικές ε, σχέσεις βοήθεια και διεύρυνση ε, και διοικητικές δεπάνες, όλες οι άλλες πολιτικές ομάδες επηρεάστηκαν από τυπικά σφάλματα. Το 2011 τα λάθη που, διαπραγμα... που διαπιστώθηκαν παρέμειναν ε, στα ίδια επίπεδα όπως και κατά τα προηγούμενα έτη. Ε, κυρίως όσον αφορά προβλήματα που δεν εμφανίζονται συχνά. Αυτό βέβαια δεν σας εκπλήσει φαντάζομαι. Θα ήταν μη ρεαλιστική η προσδοκία να υπάρξει ουσιαστική αλλαγή. Οι ρυθμίσεις ε, κυρίως ε, για το πώς δαπανούν τα χρήματα ε, προκαθορίζονται σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα. Και όπως και κατά τα προηγούμενα έτη το δικαστήριο διαπίστωσε ότι τα συστήματα ελέγχου δεν λειτουργούν πλήρως. Σε τομείς όπου έχουμε υψηλά επίπεδα προβλεπόμενου λάθους εισφάλματος, ε, οι αρχές των κρατών μελών θα πρέπει να δραστηριοποιηθούν για να εντοπίσουν τα λάθη και να ζητηθεί η επιστροφή τους ε, στον ε, προϋπολογισμό. Σε πάρα πολλούς τομείς όμως δεν επιτέχθηκε κάτι τέτοιο. Ένα καλό παράδειγμα είναι η περιφερειακή πολιτική. Εδώ, σε πάνω από 60% των ελεγχόμενων συναλλαγών, οι αρχές των κρατών μελών είχαν αρκετές πληροφορίες στη διάθεσή τους για να διορθώσουν τουλάχιστον κάποια σφάλματα πριν ζητήσουν ζητήσουν την επιστροφή χρημάτων από την Επιτροπή. Και αυτό το επιβεβαιώνει και ο έλεγχος ε, του Δικαστηρίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου το 2011 ο έλεγχος λοιπόν κατέδειξε ότι για να αποφευχθούν ε, δημοσιονομικές ε, διορθώσεις, τα κράτα-μέλη και οι αρμόδιες αρχές έχουν καταθέσει δηλώσεις, ε, οι οποίες δυστυχώς υποτίμησαν το επίπεδο σφάλματος, χωρίς κάποιες, κάποιους αποχρόνες λόγους. Τα αποτελέσματα του ελέγχου που διεξήγαγε άμεσα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως στον τομέα της έρευνας και άλλες εσωτερικές πολιτικές, κατέδειξαν ότι υπάρχουν παρεμφερείς ελλείψεις και άρα δηλαδή το μπορεί να επιστραφεί μόνο εάν υπάρχει και το ε, θετικό πιστοποιητικό από μια ανεξάρτητη αρχή. Σε πάνω από 80% των ε, ε, project που εξετάστηκαν από το ελεγκτικό συνέδριο διαπιστώθηκε ένα ή περισσότερα σφάλματα και σε περίπου 50% αυτών των περιπτώσεων ε, τα σφάλματα είχαν ουσιαστικές επιπτώσεις. Όλα αυτά λοιπόν τα παραδείγματα καταδεικνύουν ότι οι αρχές των κρατών μελών και οι Επιτροπή έχουν περιθώριο να βελτιώσουν τις δαπάνες. Βέβαια, ε, ίσως να υπάρχει μεγαλύτερο περιθώριο ε, απλουστεύοντας τους κανόνες. Ε, την περίοδο 7 έως 13 οι βασικοί κανόνες για την διαπάνη εκταμείευση των κοντιλίων αποφασίστηκαν από τα κράτη-μέλη. Έχουν δορθεί δηλαδή αρμοδιότητες εκείνους που διαχειρίζονται ενωσιακά προγράμματα. Έτσι λοιπόν τα κράτη-μέλη ε, πρέπει να στοχεύουν καλύτερα στη χρήση των κοινοτικών κονδυλίων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει βεβαίως να έχει την εποπτεία ε, των κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των δηλώσεων ε, η έκθεση ετήσιων, ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων υπεπραγμένων των γενικών διευθυντών μπορεί να καταδείξει ασφάλματα. Αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει την ασφάλεια ότι ε, τα, τα, τα κονδύλια που εκταμιεύονται ε, δεν έχουν σφάλματα. Εάν υπάρχει κάποια ασφάλεια θα πρέπει να πάψει η εκταμίευση κονδυλίων. Το 2011 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αύξησε τον αριθμό των επιφυλάξεων και αυτό αντικατοπτρίζει το ότι η Κομισιόν αναγνωρίζει ότι υπάρχουν υψηλοί κινδύνοι. Αυτό είναι ένα σημαντικό βήμα προ τα εμπρός. Η Επιτροπή πρέπει να συνεχίσει να ελέγχει του επικίνδυνου τομεί, να αποκτά απαραίτητε πληροφορίε για να έχει και του σωστού τους ε, δείκτες ε, ε, να υπάρχει υπάρχουν στοιχεία χωρίς λάθη. Στην ετήσια έκθεση του 2011 το λεκτικό συνέδριο κατέληξε στο ότι υπάρχει κάποια δυνατότητα σφαλμάτων. Τα περισσότερα προβλήματα εντοπίστηκαν από το ελεγκτικό συνέδριο και παρουσιάστηκαν Βεβαίω, ε, το ε, δικαστήριο, το ελεγκτικό συνέδριο με έχει διαπιστώσει βελτίωση κατά τα προηγούμενα έτη. Υπάρχει βέβαια και ένα ανώτατο όριο στις ε, βελτιώσεις που μπορούν να προκύψουν. Αξίζει λοιπόν τον κόπο να σκεφτεί κανείς κατά πόσον το πλαίσιο αυτό μπορεί πραγματικά να αποδώσει αυτά που επιθυμούν όλοι οι άμεσα ενδιαφερόμενοι. Μια θετική δήλωση αξιοπιστίας το, το δικαστήριο επισήμανε ότι όπου είναι αδύνατον να ε, υπάρχει συμβατότητα με τους κανόνες θα πρέπει να αναζητηθούν άλλες λύσεις ε, να απλουστευτούν οι κανόνες να υπάρχει αυστηρότερος έλεγχος υψηλότερο επίπεδο ε, μη συμβατότητας ή αν θέλετε να πάυσουν οι δραστηριότητες αυτή τη στιγμή συνεχίζονται οι συζητήσεις για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο 14 έως 20 και επίσης ε, θεωρούμε ότι η σχετική ομοθεσία αποτελεί μοναδική ευκαιρία. Η πρώτη επιτροπής για το πλαίσιο 14 έως 2020 ανοίγει την πόρτα ε, για να σχετίζουμε την απόδοση με τα κονδύλια. Τα κράτη-μέλη έχουν τη δυνατότητα, όχι όμως την υποχρέωση, να ε, εντάξουν όλα τα κονδύλια σε ένα λειτουργικό πρόγραμμα μέσα από τα αποκαλούμενα ε, κοινά προγράμματα δράσης. Βέβαια, όπως έχει αναφέρει ήδη το ε, ελεγκτικό συνέδριο στη γνωμοδότησή του του 2011, αυτή η πρωτοβουλία μπορεί να υλοποιηθεί μόνο στο βαθμό που αντικαθιστά το, την παραδοσιακή διαχείριση. Η κατάσταση τώρα στον τομέα της έρευνας ε, είναι παρεμφερής. Κατά τη διάρκεια του 7ου προγράμματος πλαίσιο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εισήγαγε τη δυνατότητα απλούστευσης έτσι ώστε να περιοριστεί το διοικητικό άχθος. Η πρόταση για το επόμενο πρόγραμμα πλαίσιο, Horizon 2020, κάνει ένα βήμα προς τα εμπρός και δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιούνται ε, κατά αποκοπή ποσά για το σύνολο των προγραμμάτων. Ίσως ε, αυτή είναι μια ε, ελκυστική λύση που ενδεχομένως αυτοί που ενδιαφέρουν να εκμεταλλευτούν δεν το γνωρίζουν γνωρίζουμε βέβαια αυτή τη στιγμή. Τα παραδείγματα αυτά καταδεικνύουν ότι υπάρχουν κάποιες προσπάθειες εκ μέρους Επιτροπής να απομακρυνθεί από το ισχύον σύστημα. Όμως παραμένει το ερώτημα. Τα κράτη-μέλη θα αναλάβουν τον κίνδυνο να απομακρυνθούν από το ε, κόστος της επιστροφής ε, εάν τα νέα μοντέλα παραμείνουν σε προαιρετική βάση και κυρίως ε, εάν είναι χαμηλό το ποσοστό σφάλματος. Αξιότιμα μέλη, το Κοινοβούλιο το Συμβούλιο καλούνται να αποφασίσουν για τους κανόνες που θα ισχύουν για τον κοινοτικό προπολογισμό. Όμως είναι βέβαια και η ευθύνη του ελεγκτικού συνεδρίου να καθορίσει την κατεύθυνση. Εμείς θα συνεχίσουμε να σας προσφέρουμε την αξιολόγησή μας, ε, των ε, δαπανών, πώς ακριβώς θα πρέπει να εκταμιεύονται οι δαπάνες με βάση τους κανόνες που έχετε εσείς οι ίδιοι καθορίσει. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι εδώ και ο... Ο κύριος Ότμπο, θέλετε να προσθέσετε κάτι. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Αξιότιμα μέλη της ε, Επιτροπής Ελέγχου Προπολογισμών. Κύριε Επίτροπε, χαίρομαι που είμαι εδώ για πρώτη φορά. Να σας παρουσιάσω το κεφάλαιο 10. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος. Είναι η δεύτερη φορά που το λεκτικό Συνέδριο έχει συμπεριλάβει ένα κεφάλαιο περί επιδόσεων στην ετήσια έκθεσή του. Ε, φέτος τρία διαφορετικά θέματα ε, πρώτον δηλαδή η αξιολόγηση, η έκθεση αξιολόγηση, δεύτερον ε, η ίδια αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τρίτον ε, το ελεγκτικό συνέδριο ασχολήθηκε με τις έξι ετήσιες εκθέσεις, με τι έξι εκθέσεις του 2011 για να ασχοληθεί με την ανάλυση τη Ευρωπαϊκή προστιθέμενης Αξία και τον προγραμματισμό. Όσον αφορά την έκθεση αξιολόγηση, ουσιαστικά λάβαμε όχι μόνο μία, μόνο μία έκθεση αξιολόγησης αλλά δύο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, γι' αυτό αναφέρομαι στο κεφάλαιο 10. Λάβαμε τη δεύτερη τον Νοέμβριο και... Ε, ήρθαμε σε επαφή με επιστολή με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Από καταλαβαίνω είναι σε ένα ξεχωριστό τίτλο που θα συζητηθεί αύριο στην Επιτροπή σας. Οπότε δεν θα προσθέσω τίποτε για την ώρα. Τώρα, τι συμπεριλάβαμε στο πρόγραμμα ίδιας αξιολόγησης Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εμείς ε, είπαμε ότι διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν ε, σημάδια βελτίωσης, ότι προχωρεί η διαδικασία, όμως υπάρχουν ακόμα προβλήματα συνοχής μεταξύ των στόχων και των δικτών, όπως επίσης και την ύπαρξη σημαντικών ε, ποσοτικών στόχων της προόδου που έχει σημειωθεί. Τι συμπέρανε το ελεγκτικό συνέδριο όσον αφορά το εγχείρημα Across the Board ε, για τις έξι εκθέσεις που καλύπτουν διάφορες ε, πολιτικές. Ε, υπήρξαν κάποια μαθήματα τα οποία όντως συμπεριλήφθηκαν, δηλαδή όταν υπήρχαν αξιολογήσεις που δεν είχαν ληφθεί σωστά επαρκώς, ε, προσπαθήσαμε τα ποσά αυτά να τα ε, κατευθύνουμε ε, σε πιο ευάλωτα προγράμματα. Επίσης υπάρχουν αδυναμίες που καθιστούν δύσκολο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει εκθέσεις για την αξιοποίηση των κονδυλίων. Επίσης είναι πρόκληση η αξιολόγηση της ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας της των δαπανών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς ε, επίσης ε, προτείνουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εστιάζει καλύτερα τις δραστηριότητες της σε ανάλυση αναγκών. Ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να βελτιώσουν την ποιότητα των προγραμμάτων που υποβάλλονται από τα κράτη-μέλη. Και τρίτο και τελευταίο, για την ε, περίοδο 2014 έως 2020 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να δείξει και να καταγράψει ε, όλα τα προγράμματα με ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί με ακούσατε σε αυτή την παρουσίασή μου του κεφαλαίου 10. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρο. Ε, ευχαριστώ και τα δύο μέλη του Ελεγκτικού Συνεδρίου για αυτέ τι πάρα πολύ καλέ ε, ε, παρουσιάσει και παρατηρήσει του. Θέλει ο Επίτροπο να απαντήσει και μετά θα γίνουν ερωτήσει. Παρακαλώ να σημειώσω τους συναδέλφους που θέλουν να υποβάλουν ερωτήσεις. Σημειώνω βέβαια και το όνομα του εισηγητή και τους υπολείπους. Κύριε Επίτροπο, έχετε το λόγο. Νομίζω ότι έχετε πολύ χρόνο στη διάθεσή σας για να πείτε σε λεπτομέρειες. Ε, ευχαριστώ πολύ, κύριε Ισηγητά. Αξιότιμα μέλη της Επιτροπής ε, Ελέγχου Προπολογισμών και του Ελεκτικού Συνεδρίου. Θα ήθελα να, τους να σας ευχαριστήσω για τον, εμπνευστικό σας, τον εμπνευσμένο σας λόγο. Συμφωνώ ότι χρειάζονται περισσότερες ε, δράσεις ε, και ότι πρέπει οπωσδήποτε να εφαρμοστούν χωρίς ε, καθυστέρηση. Πρέπει να πούμε επίσης ότι το τρέχον πλαίσιο δεν είναι ρεαλιστικό. Όταν ο προγραμματισμός δεν ήταν επαρκής, ήταν πολύ αόριστος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αξιοποίησε το επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο για να αντιμετωπίσει κάποιες από τις αδυναμίες. Αυτό έχει να κάνει με τη δομή των προγραμμάτων, με τους κανόνες, όπως επίσης και την αλυσίδα ε, λογοδοσίας ε, των οικονομικών ε, παικτών. Μέχρι τώρα έχουμε συνεργαστεί πολύ καλά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπως φαίνεται και αποτελέσματα, από τα αποτελέσματα ε, ε, του τελευταίου δημοσιονομικού πλαισίου. Όμως δεν έχει ολοκληρωθεί η δουλειά μας. Οι προτάσεις απλοποίησης τίθενται αμφιβόλο και από τους δύο συνομοθέτε Για τη μελλοντική γεωργική πολιτική περίπου 4.000 τροπολογίε έχουν υποβληθεί από ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οπότε με ανησυχεί ότι ο κοινό μα στόχο εξυγχρονισμού των προγραμμάτων, ε, μεγαλύτερη αποτελεσματικότητά του και απλοποίησή του ε, απειλείται. Χρειαζόμαστε την υποστήριξή σας για να διατηρήσουμε την ουσία αυτού που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βάσει των διδαγμάτων των εκθέσεων του Ελεκτικού Συνεδρίου και των συστάσεών του. Αν αντιθέτω είναι επαρκή ο προγραμματισμό, ε, αλλά η επίδοση των οικονομικών εταίρων δεν είναι ικανοποιητική, τότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί να παρεμποδίσει τα σφάλματα ή να τα διορθώσει συστηματικώ αυτή τη στιγμή στα εντοπίσει. Τα αποτελέσματα αυτής της ε, προσπάθειας είναι πολύ ουσιαστικά και θα σας το πω αυτό στη συνέχεια. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραμένει υπεύθυνη για την εκτέλεση του συνόλου του προϋπολογισμού, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να χαλαρώνουν οι υπόλοιποι οικονομικοί εταίροι και ειδικότερα οι αρχέ των κρατών μελών από την ανάληψη των δικών του ευθυνών και υποχρεώσεων, όπω αναφέρεται και στο άρθρο 317 της ε, Σε αρκετές περιπτώσεις ε, που φαίνεται ότι οι εθνικές ε, διαχειριστικές αρχές και οι αρμόδιες ελεγκτικές αρχές δεν έκαναν καλά τη δουλειά τους, έφτασαν ορισμένα ποσά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα οποία έπρεπε να από, να πληρωθούν παρά το γεγονός ότι δεν υπήρχε δικαιολογημένη βάση και ειδικότερα στην στην, στον τομέα της γεωργίας που είναι πολύ σημαντικό γιατί είναι το 80% του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Οι κανόνες επιλεξιμότητας μπορούν να μειώσουν το ποσοστό σφάλματος. Όμως, όπως είπα, αυτή η διαδικασία είναι πάρα πολύ αργή σε σχέση με τις προτάσεις των, ε, για τους νέους κανονισμούς. Σήμερα, όπου έχουν γίνει απλοποιήσεις στο τρέχον νομοθετικό πλαίσιο δεν χρησιμοποιούνται από τα κράτη-μέλη και το γεγονός ότι έγιναν 13 αξιολογήσεις από ανεξάρτητα τα όργανα ελέγχου δείχνει ότι έχουν μικρή όρεξη οι εθνικές αρχές για τη χρήση αυτών των, αξιοποιήσεων, των, αξιο, των απλοποιήσεων επιτόπου ε, σε σχέση με τους δικαιούχους, ε, ε, με την καλύτερη πρόσβαση στη χρηματοδότηση και την μείωση του ποσοστού σφάλματος θα γνωρίζετε ότι οι κανόνες επιλεξικότητας και συνοχής ε, ορίζονται σε εθνικό επίπεδο. Για το 2011, 86% του ποσοστού σφάλματος για τα κοινωνικά ταμεία είχε να κάνει με, την εθνική, με τους εθνικούς κανόνες επιλεξιμότητας. Οπότε, παρά την ε, συνεχή έκκληση από την πλευρά τη Επιτροπής, ε, δεν φαίνεται να προβαίνουν σε ιδιαίτερη απλοποίηση σε εθνικό επίπεδο. Και σύμφωνο βέβαια ότι δεν είναι καλό να αλλάζουμε συχνά κανόνες. Πάντως το νέο ε, δημοσιονομικό πλαίσιο, πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, δίνει αυτή τη δυνατότητα για 7 χρόνια. Και εδώ η Κομισιόν θα ε, θέλει να έχει δική σας υποστήριξη. Όσον αφορά την κοινή διαχείριση και την απόδοση των εθνικών αρχών, όπως επίσης και τον σχεδιασμό των κανόνων επιλεξιμότητας, είναι καθοριστική σημασία να περιοριστεί το υπολοιπόμενος, κίνδυνο σφάλματο. Και θέλω να πω ότι οι εθνικές αρχές ε, ε, όταν βρίσκονται σε σύγκρουση με το ελεγκτικό συνεδρίο, αυτό είναι καθοριστικό για πολλούς λόγους. Πρώτον, μπορούν όσοι άμεσα εμπλέκονται να προσφέρουν τις απαραίτητες εξηγήσει για να αξιολογηθεί η κατάσταση. Επίσης, οι εθνικές αρχές, οι εμπλεκόμενες, είναι υποχρεωμένες να ελέγξουν προσεκτικά τα πορίσματα του ελέγχου και επίσης και να διευκρινίσουν την πηγή. Άρα δηλαδή πρόκειται για μια αμφίδρομη διαδικασία η οποία μπορεί να ε, βελτιώσει την κατάσταση επιτόπου. Και αυτό ισχύει για όλα τα προγράμματα του κοινή διαχείριση, συμπεριλαμβάνει και τη γεωργική και τη περιφερειακή ανάπτυξη. Και τώρα θα ήθελα να σχολιάσω λιγάκι τα βασικά θέματα και τι ερωτήσει που ετέθησαν από την Επιτροπή σε προηγούμενε ακροάσει και σε συζητήσει για την απαλλαγή. Πρώτον, όσον αφορά τη δυνατότητα διόρθωση του υφιστάμενου συστήματο ελέγχου. Το Νοέμβριο του προηγούμενου έτου σα εξήγησα ότι το σύστημα ελέγχου οδήγησε στο να ανακτηθούν και να διορθωθούν 1,84 δισεκατομμύρια ευρώ το 2011. Είναι ένα τεράστιο ποσό που αναλογεί στο 1,4 όλων των πληρωμών που έγιναν το 2011. Ακόμα και αν το ποσό αυτό αφορά τις πληρωμές προηγούμενων ετών από την προοπτική προστασία του Ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού το 2011 αξίζει τον κόπο να το σκεφτεί κανείς μέσα σε ένα ευρύτερο πλήρωμα Τόσο οι διορθώσεις όσο και οι ανακτήσεις ε, καταγράφονται στους ετήσιους ε, λογαριασμούς Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, για πέμπτο συναπτό έτος. Βέβαια δεν περιλαμβάνουν στοιχεία για δημοσιονομικές διορθώσεις και ανακτήσεις που έγιναν από τα ίδια τα κρατημέλη διότι μέχρι τώρα τα στοιχεία δεν ήταν αξιόπιστα και υπάρχει ο κίνδυνος του διπλού υπολογισμού την, ε, στους επόμενους λογαριασμούς οι αρμόδιοι θα διασφαλίσουν την ποιότητα των δεδομένων έτσι ώστε να μπορεί κανείς να τα χρησιμοποιήσει στους λογαριασμούς. Και επιπλέον η αναφορά προληπτικών και διορθωτικών μέτρων παρουσιάστηκαν στο σημείο με υπαριθμών 6 των λογαριασμών και αυτά όλα θα είναι πολύ πιο φιλικά για το χρήστη το 2012. Δεύτερον, θα ήθελα τώρα να αναφερθώ λιγάκι στους ε, τομείς πολιτικής υποκοινή διαχείριση. Όσον αφορά την γεωργική ανάπτυξη. Η Κομισιόν έχει καθορίσει πρόγραμμα δράσης για να εξετάσει ε, την κατάσταση που εντόπισε το ελεγκτικό συνέδριο, να εντοπίσει τις αδυναμίες και να λάβει διορθωτικά μέτρα. Πιο συγκεκριμένα, η Κομισιόν έχει ενημερώσει τις διοικήσεις όλων των κρατών μελών σε διάφορες περιπτώσεις σχετικά με τα αίτια των σφαλμάτων και το τι είδου διορθωτικές πράξεις μπορούν να αναλυφθούν. Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Γεωργικής Ανάπτυξης θα βοηθήσει στο να υπάρχει καλύτερη συνειδητοποίηση για τα θέματα αυτά. Η κατάρτιση και η καλύτερη ενημέρωση έχουν προσφερθεί στους ε, δικαιούχους. Η Γενική Διεύθυνση Άγκρη έχει ε, προσαρμόσει το πρόγραμμα ελέγχου της ε, το 2011 και έχουν επισημανθεί στα κράτη-μέλη οι ψηλότεροι κίνδυνοι που υφίστανται. Τέλος, ε, το ε, προσωπικό της ομάδας ελέγχου της γεωργικής ανάπτυξης θα ενισχυθεί ως προς το μέλλον. Και εκτός από τα πλουστευμένα προγράμματα πληρωμών έχουν ε, εξεταστεί και άλλα μέτρα, όπως ας πούμε υποχρέωση στο μέλλον να υποβάλλονται προγράμματα γεωργικής ανάπτυξης ε, πριν από την έγκριση της ε, Κομισιόν ε, σε αρμόδιες υπηρεσίες των κρατών μελών, έτσι ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος σφάλματος. Ως προς την πολιτική συνοχή. Η κατάσταση βελτιώθηκε ουσιαστικά πέρυσι και θεωρώ ότι θα υπάρξει περαιτέρω βελτίωση μόλις αρχίσουν να, να γίνονται αισθητέ οι επιπτώσεις από τον δημοσιονομικό κανονισμό. Σε αυτή την τρέχουσα περίοδο ε, οι εθνικές αρχές ε, ελέγχουν ε, τα προγράμματα και ζητούν ε, δημοσιονομικές διορθώσεις. Τα κρατημέλη τώρα πλέον είναι υποχρεωμένα να αναφέρουν ε, τις πράξεις τους και να διορθώνουν τις ε, αδυναμίες. Στην περίπτωση που κρίνεται μη επαρκής η πρόοδος, λαμβάνονται προληπτικά μέτρα όπως διαδικασία προκατακτική διαδικασία αναστολής. Ο στόχος δεν είναι να περιστούν οι πληρωμές, αλλά να διασφαλιστεί ότι και οι εθνικές αρχές εφαρμόζουν τις ε, αρχές της υγιούς, της χρηστής οικονομικής διαχείρισης. Επιπλέον, η Γενική Διεύθυνση Ρίτζο και Απασχόλησης ε, είναι εκείνε που θέλουν να εστιάσουν την προσοχή τους στα πιο επικίνδυνα προγράμματα. Οι αρχές των κρατών μελών πρέπει να στηριχθούν στη βελτίωση των δικών τους των προγραμμάτων κατάρτισης για να διασφαλίσουν την εφαρμογή των εθνικών κανονισμών. Η Γενική Διεύθυνση Ρίτζο έχει ιδρύσει ένα κέντρο ε, με ακριβώς αυτό το σκοπό το στόχο. Για την αμέσως επόμενη περίοδο προβλέπεται η εισαγωγή μιας ε, δήλωσης διαχείρισης για όλες ε, τις ε, δαπάνες που πραγματοποιούνται υπό κοινή διαχείριση. Έτσι λοιπόν αυτό θα συμβάλλει στην διαδικασία πιστοποίησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και από τη στιγμή που θα εφαρμόζεται πλήρως το σύστημα αυτό και θα μπορεί κανείς να αξιολογήσει τις επιπτώσεις. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα κάνει το δεύτερο βήμα και θα στηρίξει ανεπιφύλακτα σε πολιτικό επίπεδο αυτή τη νέα διαδικασία απόδοσης λογαριασμών που θα εισάγουν τα κράτη-μέλη. Πάμε τώρα στην έρευνα. Ένας τομέας όπου η Επιτροπή ε, θεωρεί ότι υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό σφάλματος. Η αύξηση του ποσοστού σφάλματος ε, ε, πέρυσι αφορά κυρίως ε, τις διαδικασίες αναφοράς και επαλήθευσης. Οι περισσότεροι έλεγχοι αφορούσαν το διοικητικό άχθος με κίνδυνο τα προγράμματα έρευνας και καινοτομία στην Ευρώπη να μην είναι πλέον ελκυστικά. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να υπάρχει μια καλή ισορροπία ανάμεσα στην εμπιστοσύνη και τους ελέγχους, όπως ζητήθηκε από την έκθεση Μέρκης ε, που εγκρίθηκε το Μάιο του 2011. Εδώ λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναθεωρεί τους ελέγχους της, εστιάζει περισσότερο σε επικίνδυνες συναλλαγές και στην περίπτωση να διαπραχθούν απάτες. Ε, ένα σχετικό ερωτηματολόγιο θα απαντήσει ε, τις ερωτήσεις των ε, ενδιαφερόμενων με συντονισμένο τρόπο. Αυτό θα προσφέρει την δυνατότητα να συμμετέχουν και οι άμεσα ενδιαφερόμενοι και οι ελεγκτές. Τώρα, ε, feedback θα υπάρχει άμεσα από τις ε, γενικές διευθύνσεις ε, προς ανεξάρτητους ελεγκτές, οι οποίοι όμως δεν, προσφέρουν, δεν θα προσφέρουν ικανοποιητική ποιότητα. Αυτοί θα κληθούν από την Επιτροπή σε ένα σχετικό σεμινάριο. Θα υπάρχουν ειδικά προγράμματα εκπαίδευσης για αυτούς. Στην περίπτωση που ε, δεν εντοπίζονται έγκαιρα οι αδυναμίες της εκθέσεις τους, η Κομισιόν θα καλέσει ε, τους άμεσα υποφελούμενους να καταγγείλουν τις συμβάσεις αυτών των ελεγκτών. Στο μέλλον, η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα περιλαμβάνει και τις ε, βέλτιστες δυνατότητες δαπανών. Με τον τρόπο αυτό ελπίζουμε ότι θα μπορεί κανείς να επιτύχει καλύτερα τους στόχους. Είναι λοιπόν καθοριστική σημασία ε, η πρώτη Επιτροπή να στηριχθεί από το Κοινοβούλιο γιατί όλους μας μας ενδιαφέρει να προχωρήσουμε σε ε, χρηστή διαχείριση. Και θέλω να υπενθυμίσω ότι εσείς ε, έχετε κάνει κάποιες τροπολογίες οι οποίες όμως ενδεχομένως να θέσουν σε κίνδυνο τα προγράμματα έρευνας και καινοτομία. Τέταρτον, τώρα θα πάω στην σε θέματα προϋπολογισμού. Εκεί δηλαδή όπου ε, μπορούν να ε, λειτουργήσουν ε, συνεργασίες με τις κυβερνήσεις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί συνεχώς να επιτύχει βελτίωση στον έλεγχο αυτού του τομέα δαπανών, έτσι ώστε η βοήθεια να μπορεί να χρησιμοποιείται αποτελεσματικότερα. Μέχρι το 2013 ελπίζουμε ότι θα υπάρξει περαιτέρω βελτίωση με βάση τις συστάσεις του ελεγκτικού συνεδρίου. Πρόκειται κυρίως για το ε, για τη διαχείριση, για την ομάδα στήριξης του προϋπολογισμού, κυρίως όλα αυτά σε ανώτατο πολιτικό επίπεδο. Πρέπει να υπάρχουν πιο αυστηροί έλεγχοι και αξιολογήσεις. Τέλος, η αξιολόγηση των κοινοτικών προγραμμάτων για την απόδοσή τους, ε, αυτό πρέπει να γίνει για να υπάρχει ε, διασφάλιση της αποτελεσματικότητας. Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, προσβλέπουν σε πραγματικά ωφέλη και προστιθέμενη αξία από τις δραστηριότητές τους. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς ενισχύουμε το σύστημά μας έτσι ώστε να εξετάζουμε το θέμα της εκτέλεσης του προϋπολογισμού σε τακτά χρονικά διαστήματα. Με την τελευταία έκθεση αξιολόγησης ε, μπορεί κανείς να έχει περισσότερα στοιχεία για την έκθεση αξιολόγηση επιτροπής. Η Επιτροπή θεωρεί, όπως και το ελεγκτικό συνέδριο εξάλλου, ότι ε, πρέπει να ε, συμφωνούν με την αρχή απαλλαγής για το πώς ακριβώς θα συντάσσεται η έκθεση και τι είδους πληροφορίες θα δίδονται. Όπως και το δικαστήριο και εγώ πιστεύω ότι πρέπει να προχωρήσουμε ε, σε προγράμματα που έχουν, είναι στοχευμένα στο στόχο και από τα οποία προσβλ... μπορεί να περιμένει προστιθέμενη αξία. Γνωρίζω ότι υπάρχει πλέον μια μετακίνηση από ε, το input σε impact και ε, θεωρώ επίσης ε, ότι και αυτά τα δύο σχετίζονται άμεσα με τη διαδικασία απλούστευσης. Η επιτυχία θα εξαρτηθεί από τη βούληση των συνομοθετών όλα αυτά να τα καταστήσουν εφικτά. Αγαπητά μέλη, θα ήθελα να κλείσω τη σύντομη παρέμβασή μου διαβεβαιώνοντάς σας ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη μάθει το μάθημά της από αυτή τη διαδικασία απαλλαγής και θα προσπαθήσει από κοινού με άλλους ε, δημοσιονομικούς εταίρους και με εσά να συνεργαστεί. Ε, μπορώ να σας διαβεβαιώσω λοιπόν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ανοιχτή σε πρωτοβουλίες που θα οδηγήσουν σε βελτιωμένη δημοσιονομική διαχείριση ε, και σε δράσεις ε, που θα πρέπει να αναλυφθούν με βάση τις συστάσεις που έχουν δημοσιευτεί στην ετήσια έκθεση η αέναη βελτίωση είναι ένας στόχος που δεν, δεν μπορεί να τον πετύχει μόνη της η Κομισιόν, μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από ομαδική εργασία με την βοήθεια των συνομοθετών, των αρχών προπολογισμού και απαλλαγή. Και εκεί όλοι οι ελεγκτές και όλοι οι οικονομικοί παράγοντες μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο. Σα ευχαριστώ για την προσοχή σας. Als rapporteur. Θα δώσουμε το λόγο στον εισηγητή. Κύριε Πρόεδρε, ε, Μπάρτ, ε, σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Επίτροπε, καταρχήν σας ευχαριστώ για το ότι απαντήσατε στις ερωτήσεις ε, εκτενώς και σας ευχαριστώ πολύ και για όλα αυτά που μας είπατε. Αυτά που μας είπατε βασίζονται σε μια σε την επικοινωνία που είχαμε εμείς μεταξύ μας όπου κατά κάποιον τρόπο ε, είχαμε συμφωνήσει που θα βασίζεται, που θα εντράζεται η ε, έκθεση απαλλαγής. Δεν μπορώ να κάνω ερωτήσεις γιατί έχετε ήδη δώσει όλες τις απαντήσεις. Εκείνο που θέλω να κάνω είναι να επισημάνω κάποια θέματα που μπορεί να προκαλέσουν αντιδράσεις. Κοιτάξτε, εσείς δεν είσαστε μόνο αρμόδιοι για την απαλλαγή, αλλά και για τα δασμολογικά και για τα έσοδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέχρι τώρα Αυτά δεν τα προβάλαμε ιδιαίτερα στις εκθέσεις απαλλαγής, γιατί το ελεγκτικό συνέδριο απλά ε, ελέγχει κατά πόσον καταγράφονται και καταχωρίζονται σωστά τα έσοδα. Εγώ λοιπόν θεωρώ ότι δεν πρέπει να εξτάζουμε μόνο την καταγραφή, αλλά και το περιεχόμενο των εσόδων. Και μακροπρόθεσμα να δούμε πώς μπορούμε να διαχωρίσουμε το τι πρέπει να γίνει μακροπρόθεσμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση από την απαλλαγή. Έχουμε λοιπόν το θέμα ε, του δημοσιονομικού πλαισίου από το 2014. Αυτό είναι ε, ένα επίμαχο θέμα και γι' αυτό το λόγο πρέπει να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα έσοδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως στον τομέα που μας αφορά. Ε, παρότι ε, δεν ασχολείται το ελεγκτικό συνέδριο με το θέμα αυτό στην ετήσια έκθεσή του, γενικά αναφέρεται βέβαια σε αυτό και μας επισημαίνει ε, το ελεγκτικό συνέδριο πάντα ότι υπάρχουν δυνατότητες ε, βελτίωσης κυρίως στον τομέα των τελωνίων και των δασμών. Εμείς λοιπόν πράγματι μεταβήκαμε επί τόπου, είδαμε λιγάκι το πώς συγκεντρώνονται τα δασμολογικά στοιχεία στην ε, Αμβέρσα και στο Ρότερνταμ και θέλω να σας πω ότι τα προγράμματα των ε, κρατών μελών αυτά που έχουν κυρίως ε, στόχο της τα δασμολογικά έσοδα, σε αυτό τον τομέα τα κράτη-μέλη είναι πολύ αναβλητικά. Και γιατί, διότι λένε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι εκείνη που πρέπει να ασχολείται με την ε, ίσπραξη κονδυλίων. Βεβαίως όλο αυτό είναι ιδιαίτερα χρονοβόρο. Τα κράτη-μέλη ε, το νέο δασμολογικό κανονισμό να μην τον εισάγουν παρά μόνο το 2020. Και αυτό εμάς δεν μας ικανοποιεί. Άρα δηλαδή η πρώτη μου παράκληση είναι η εξή. Εσείς τι πιστεύετε για όλα αυτά και τι σκοπεύετε να κάνετε τόσο για τα έσοδα από το ΦΠΑ όσο και για τα έσοδα από τους δασμούς. Πώς αξιολογείτε τις επικείμενες εξελίξεις. Νομίζω ότι αυτό για το θέμα της απαλλαγής μπορεί να μην είναι καθοριστική σημασίας, αλλά είναι σημαντικό για το πώς θα κάνουμε τη δουλειά μας και πώς ε, μπορούμε να αξιολογήσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το δεύτερο θέμα που θέλω να δείξω αφορά εσάς επειδή είστε ο αρμόδιος επίτροπος για την απαλλαγή. Θα κάνω μια φιλοσοφική ερώτηση. Κοιτάξτε δηλαδή να δούμε πώς δουλεύει η Επιτροπή, ε, το πώς κάνει τι αναλύσεις. Αυτά είναι σημαντικά. Γιατί τι γίνεται, συμβαίνει το εξή. Θα τα πω κάπως αλλιώς τώρα, θα τα πιάσω από άλλη πλευρά. Αυτά οι σκέψεις που μας οδηγούν στην απαλλαγή ε, βασίζονται σε δύο πράγματα στην έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου, στην ειδική έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου και βεβαίως και στα έγγραφα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και έτσι έχουμε πρόβλημα ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όχι μόνο στην ερμηνεία του ποσοστού σφάλματος αλλά και στη σημασία αυτού. Έχουμε δηλαδή το ελεγκτικό συνέδριο το οποίο αξιολογεί τα σφάλματα με βάση το ένα, την κλίμακα 1% και έχουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία ασχολείται με σφάλματα μόνο εφόσον αυτά συνδέονται με συγκεκριμένα ποσά. Πρέπει λοιπόν να γνωρίζουμε ότι εμείς εδώ κάνουμε μια δουλειά που ενδιαφέρει πάρα πολύ τον Ευρωπαίο πολίτη, διότι πιστεύουν ότι με τη δική μας δουλειά ε, προστατεύουμε καλύτερα τα χρήματα του φορολογούμενου. Άρα δηλαδή καλούμεθα να απαντήσουμε στο ερώτημα ποιο είναι το ποσό εκείνο το οποίο τελικά μπορεί να αντιμετωπίσει προβλήματα στον ευρωπαϊκό, στον κοινοτικό προϋπολογισμό. Έχουμε λοιπόν το ποσοστό λάθους. Το ποσοστό αυτό λάθος βασίζεται σε δειγματοληπτικές έρευνες, μεταφέρεται αυτό στο σύνολο του προϋπολογισμού και από εκεί εξάγονται συμπεράσματα. Αυτό όμως δεν είναι σοβαρό. Αν δούμε λιγάκι ποια είναι η πραγματική οικονομική ζημιά τότε και τα στοιχεία που μας δίνει το ελεγκτικό συνέδριο δεν βοηθούν γιατί είναι άκαμπτα, είναι πάρα πολύ άκαμπτα. Από την άλλη βέβαια έχουμε τις, ε, τους κανόνες ε, που ε, προβλέπει η συνθήκη σε σχέση με τη μέθοδο της δήλωσης αξιοπιστίας και έχουμε και ένα ποσοστό ε, σφάλματος, κυρίως ε, του ε, σημαντικού σφάλματος. Ξέρετε κάτι, αυτό είναι συσήφιο έργο. Γιατί τι γίνεται, υπάρχουν λόγοι που οδηγούν στο να πρέπει να αλλάξει αυτή η μέθοδος. Η συζήτηση βέβαια δεν πρέπει να ξεφύγει τελείως, αλλά εκείνο που αντιμετωπίζουμε είναι να υπάρχει τεχνητή διόγκωση του σφάλματος, του ποσοστού σφάλματος, διότι τροποποιείται ο αριθμός των σφαλμάτων, λέει ο μιλητής. Διογκούται το κατόφλι και αυτή η διόγκωση προκύπτει από μια τεχνική βάση υπολογισμού. Αγαπητοί συνάδελφοι, χαίρομαι που θα κάνουμε την κουβέντα αυτή. Ε, θα προσπαθήσουμε πραγματικά να ερμηνεύσουμε σωστά αυτούς τους αριθμούς. Αλλά ξέρετε, να σας πω το εξής... Ε, εμείς εδώ τα καταλαβαίνουμε, οι άλλοι συνάδελφοι πολιτικές ομάδες δεν τα καταλαβαίνουν και θα πρέπει να τους βοηθήσουμε. Και το θέμα είναι πότε θα μπορέσουμε επιτέλους ε, να φτάσουμε ε, σε μια πραγματική δήλωση αξιοπιστίας χωρίς ποσοστά ασφάλματος. Σας είπα, εδώ αισθάνομαι σαν το σύσυφο πάω προς τα πάνω, ανεβαίνω, ανεβαίνω, ανεβαίνω και μόλις φτάσω και νιώθω ότι μείωσα επιτέλους το ποσοστό σφάλματος, άντε τώρα πάλι από την αρχή, αλλαγές, αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού και τι γίνεται η μπάλα αυτή που έχω με κόπο ανεβάσει στην κορυφή πέφτει και με καταπλακώνει. Βεβαίω ε, η Κομισιόν μπορεί να μου πει και τι γκρινιάζει. Ε, ο Σύσυφο ήταν ευτυχή. Μια χαρά ήταν. Αλλά εμεί δεν μπορούμε να αντιμετωπίζουμε με τον τρόπο αυτό τη δουλειά μα. Και θα πρέπει λοιπόν να δούμε πώς επιτέλους με αυτή τη μέθοδο αξιοπιστίας μπορούμε να σημειώσουμε ε, πρόοδο μπορούμε βέβαια να κάνουμε αυτό που προτείνουν οι Ευρωπαίοι συντηρητικοί. Που να λένε αφού δεν υπάρχει πραγματική δήλωση αξιοπιστίας να μην δώσουμε απαλλαγή και να προκύψει χάος. Ε, δεν είναι και αυτό λύση. Υπάρχουν κάποιοι τομείς που τα πράγματα πάνε αρκετά καλά. Ακούω ας πούμε στη Γενική Διεύθυνση απασχόλησης ότι υπάρχουν αυτές οι περίφημες τριμερείς ε, συναντήσεις και συζητήσεις όπου οι Κομισιόν οι Εθνικές Αρχές και οι τελικοί αποδέκτες συζητάνε για το πώς είναι δυνατόν να περιοριστεί ε, το ποσοστό σφάλματος. Και για δες, φτάσαμε περίπου σε ένα αποδεκτό κατόφλι για του χρόνου στο περίπου 2%, άρα δηλαδή Τελικά ο Σύσυφος μπορεί να μην ήταν και τόσο δυστυχής, λέει ο μιλητής. Το θέμα είναι το εξή. Εμεί ω Επιτροπή Ελέγχου Προπολογισμών βρισκόμαστε σε μια δύσκολη κατάσταση γιατί έχουμε δύο μεθόδου υπολογισμού του σφάλματο. Η μία μέθοδο αφορά την Κομισιόν και η άλλη μέθοδο αφορά το ελεγκτικό συνέδριο. Εμεί τώρα δεν θέλουμε να μπούμε στη μέση και να παίξουμε το διαιτητή και να πούμε έχει ο ένα ή ο άλλο δίκιο. Εμά. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να εξευρεθεί μια πολιτική λύση. Εμένα με ενδιαφέρει ε, να μου πείτε ποιες είναι οι σκέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Βεβαίω υπάρχει ένα θέμα που θα μπορούσε να μας βοηθήσει λιγάκι να βγούμε από το πρόβλημα. Ξέρετε ποιο, το να γνωρίζουμε τελικά ποια είναι τα κονδύλια εκείνα που εισπράττει η Επιτροπή. Όταν την πρώτη φορά συζητήσαμε για το ποσοστό σφάλματος, τότε ο καθηγητής κύριος Μπονίτσι, ε, που συμμετέχει στο, ε, είναι μέλος του ελεγκτικού συνεδρίου, υπάρχουν δύο μέθοδοι. Ή θα αυξήσουμε τους ελέγχους, για να περιοριστεί το ποσοστό σφάλματος, άρα η compliance, η συμβατότητα ε, θα είναι πιο αυστηρή, ή θα διορθώσουμε τα λάθη. Αυτή βέβαια είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα προσέγγιση. Το ελεγκτικό συνέδριο τοποθετείται επ' αυτού. Πάντως ε, τα κονδύλια που έχουν εισπραχθεί θα πρέπει να συσχετιστούν με χρήσεις, με συγκεκριμένα δημοσιονομικά έτη ε, και βεβαίως υπάρχουν κάποιοι σχετικοί δείκτες. Αυτή τη στιγμή η τεκμηρίωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν είναι τέτοια έτσι ώστε να έχουμε στα χέρια μας ένα έγγραφο όπου να μπορεί κανείς να δει ποια είναι τα ποσά που εισπράχτηκαν σε μία και μόνο χρονιά. Και δεύτερον, δεν μπορεί κανείς να δει σε ποια δημοσιονομική χρήση αναφέρονται τα ποσά αυτά. Αν υπήρχε αυτό, θα μπορούσε να μας βοηθήσει. Γιατί τώρα, αυτή τη στιγμή, σας είπα, ε, βλέπουμε ότι υπάρχει ένα ποστό σφάλματος που δεν μπορούμε να το ελέγξουμε. Μετά εισπράττονται χρήματα που ε, δεν μπορεί να εντοπίσει κομισιόν. Κατά την εφαρμογή του προπολογισμού, όπως σας είπα, υπάρχει ένα ποσοστό σφάλματος και αυτό που ενδιαφέρει είναι να δούμε η Κομισιόν από τη στιγμή που εντοπίσει ένα σφάλμα πόσο πίσω μπορεί να πάει και να ζητήσει την ανάκτηση κονδυλίων. Δηλαδή, ας υποθέσουμε ότι στο χρονικό διάστημα 2000 μέχρι 2006, σε αυτή την ε, εμπορική περίοδο, είχαμε κατέτος ποσοστά σφάλματος, όπως διαπίστωσε εξάλλου και το ελεγκτικό συνέδριο, και αυτά θα συσχετιστούν με αιτήματα για ανάκτηση ποσών. Ε, που τι θα σήμαινε αυτό, θα περνάγαμε το μήνυμα προς τα έξω ότι είναι εντάξει, γίνανε λάθη, αλλά ζητήσαμε πίσω τα χρήματα. Και αυτό θα ήταν μια πολύ σημαντική, ένα πολύ σημαντικό πολιτικό μήνυμα. Πρέπει να σας πω ότι με μεγάλη μου χαρά άκουσα ότι στα σημεία όπου εντοπίζεται ουσιαστική επιδείνωση του ποσοστού σφάλματος όπου το ελεγκτικό συνέδριο εντοπίζει επιδείνωση του ποσοστού σφάλματος, εκεί το ελεγκτικό συνέδριο καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει πρωτοβουλίες για βελτίωση. Αυτό μάλιστα εγώ λέω να το απαιτήσετε. Μέχρι το Μάιο θα ήθελα να δω τι βήματα θα κάνει η Κομισιόν στους τρεις αυτούς τομείς, κυρίως όσον αφορά το σημαντικό ποσοστό λάθους. Τι προτίθεστε να κάνετε, έτσι ώστε να περιορίσετε το ποσοστό σφάλματος. Στη τελική ανάλυση, ειδικά στην περιφερειακή πολιτική, εμένα με ενδιαφέρουν δύο θέματα, δεν είπατε τίποτα από αυτό, αλλά μπορείτε να επανέλθετε. Το ένα θέμα που με ενδιαφέρει και νομίζω ότι ομιλώ εκ μέρου εξ του συνόλου της Επιτροπής είναι ότι δεν είμαστε ικανοποιημένοι που υπάρχουν αναδρομικά προγράμματα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν προκύπτει προστέμενη αξία από τέτοιου είδους αναδρομικά προγράμματα. Όταν υπάρχουν προγράμματα ε, όπου εκ των υστέρων επικαλείται ο ενδιαφερόμενος την ευρωπαϊκή βοήθεια, αυτά δεν είναι επικοδομητικά. Αυτά τα αναδρομικά προγράμματα, σας λέω, ή τα προγράμματα που εκ των υστέρων ζητούν την κοινοτική βοήθεια, εκεί τα ποσοστά ασφάλματος είναι αρκετά υψηλά. Και αν τα ανακαλέσουμε, τότε πραγματικά αυτό θα πονέσει τα κράτη-μέλη και εγώ θα χαρώ πάρα πολύ. Γνωρίζω από τη Γενική Διεύθυνση Ρέγκιο ότι όσον αφορά αυτά τα αναδρομικά προγράμματα επιθυμούν να υπάρχει αυστηρότερη διαχείριση. Και αν αυτό το ζητήσουμε εμείς ως Κοινοβούλιο, νομίζω θα προχωρήσουμε πάρα πολύ. Και θεωρώ ότι θα μπορέσουμε ε, να τα πετύχουμε όλα αυτά με τη μεταρρύθμιση ε, του ε, Ταμείου Συνοχής. Και το δεύτερο θέμα που θέλω να δείξω είναι οι καθαρές διορθώσεις. Και εδώ συνεχίζω κάτι που το είπε ήδη ο προκάτοχός μου, ο κύριος Φιέλνερ. Δηλαδή, τα κράτη-μέλη μπορούν να μεταφέρουν κονδύλια από ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα σε ένα άλλο, εάν το αρχικό παρουσιάζει λάθη. Εγώ το βρίσκω αυτό σωστό. Ο κ. Φιέλνερ έλεγε καλύτερα να ε, διαγραφεί πλήρως αυτό το πρόγραμμα. Όχι, δεν είναι σωστό. Εγώ θεωρώ ότι να, αυτό είναι ένα κίνητρο να βελτιωθούν τα κράτη-μέλη. Καλύτερου ελέγχου να διεξάγουν. Αν όμω δεν βελτιωθούν, για μένα ας πούμε, αυτό είναι πολύ σημαντικό, ε, χάρη, ε, υπήρξε ένα έτο όπου τα τα κράτη-μέλη διαπίστωσαν ένα τεράστιο αριθμό ε, σφαλμάτων. Αν βέβαια τα κράτη-μέλη δεν διορθώνουν τα σφάλματά του, τότε πράγματι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ε, ανακαλεί, να διεκδικεί την επιστροφή κονδυλίων. Θεωρώ ότι αυτό στο κάτω-κάτω προστατεύει τα χρήματα του Ευρωπαίου φορολογούμενου. Θέλω να αφήσω το λόγο και σε άλλους συναδέλφους. Εγώ θέλω να πω και κάτι άλλο για την performance evaluation, αλλά εν πάση περιπτώσει ας το πει κύριος Chris Davis. Στο σημείο αυτό κλείνω την παρέμβασή μου. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον εισηγητή και ε, θα ήθελα να μου επιτρέψετε ε, να σας ε, καλωσορίσω. Αναφερθήκατε στον Καμού, στον Αλμπέρ Καμού και Όσον αφορά όμως ε, τις καιρικές συνθήκες, εγώ περισσότερο θυμάμαι τον Κάφκα. Ο Καμίου βέβαια είπε ότι μπορεί κανείς να ξεπεράσει την περιφρόνηση παραπέμποντας ο Καμίου στον Σύσυφο. Έχω λοιπόν εδώ ένα πολύ μεγάλο κατάλογο μιλητών. Τον πρώτο, ο πρώτος που έχει δει στο λόγο είναι ο κύριος Πίπερ. Κύριε Πρόεδρε, Κύριε Επίτροπε, συνάδελφε Γκάια, βεβαίω ε, το να μιλήσει κανείς μετά από εσά, ε, αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εσείς τα είπατε όλα σχεδόν, τα εξαντλήσατε. Αλλά εγώ παρόλα αυτά θα προσπαθήσω να αναφερθώ σε κάποια θέματα που ελέγχθησαν. Κοιτάξτε, θέλω να πω το εξή. Παρότι έχουμε, έχουν ε, ε, γίνει αυστηρότερη ελέγχοι, παρόλα αυτά διαπιστώνεται ένα υψηλό ποσοστό σφάλματος. Και διαρωτώ με, σε αυτό το σύστημα ελέγχου, μα τι είναι εκείνο που δεν πάει καλά. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μήπως ε, κάνει πολύ εύκολη τη ζωή της και λέει ότι σε τελική ανάλυση την ευθύνη την φέρουν τα κράτη-μέλη γιατί έχουν τις απαραίτητες πληροφορίες. Όχι κύριε Επίτροπε, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ε, η τελευταία, η ο τελικός λόγος ε, βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή που εκείνη είναι ο θεματοφύλακας των συνθήκων. Εγώ λοιπόν πιστεύω ότι πρέπει να σκεφτούμε πώς μπορούμε ως Επιτροπή ε, να ασκούμε μεγαλύτερο έλεγχο και εσείς δηλαδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πάντα σε σχέση με τους ελέγχους διότι με βάση αυτά που ακούσαμε από το ελεγκτικό συνέδριο υπάρχουν ακόμα μεγάλα ποσοστά σφάλματος. Αυτό ήταν το πρώτο ερώτημα και το δεύτερο ερώτημα που θέλω να κάνω είναι το εξή. Ε, έχει άμεση σχέση με αυτά που είπε ο κύριος Γκάια. Διότι πράγματι υπάρχουν πολιτικοί που βρίσκονται εδώ στο Κοινοβούλιο και είναι πέντε, άλλοι πάλι αν είναι τυχεροί είναι και δέκα χρόνια. Και όλοι αυτοί εκνευρίζονται πάρα πολύ όταν δεν μπορεί να γίνει η σύγκριση με παλαιότερα τη σύγκριση σε ποσοστά λάθους, σε εισπραχθέντα ποσά. Δεν υπάρχει καμία δυνατότητα σύγκρισης. Ε, έτσι λοιπόν αυτό μας κόβει τα χέρια. Δεν έχουμε ουσιαστικά καμία δυνατότητα να φτάσουμε στην ουσία του προβλήματος. Και έτσι λοιπόν εσείς ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εμείς ως Κοινοβούλιο, αν θέλουμε να διεκδικούμε την εμπιστοσύνη, τότε πρέπει να διεκδικήσουμε τη συγκρισιμότητα. Να μπορεί κανείς να συγκρίνει με παλαιότερα έτη για να διαπιστώσει τι βελτιώθηκε και τι επιδεινώθηκε. Και νομίζω ότι αυτό ήθελε να πει και ο συνάδελφος κ. Γκάιερ, και για αυτό το θέμα θα ήθελα να σας στηρίξω ανεπιφύλακτα έτσι ώστε να βρούμε από κοινού μία σωστή μέθοδο. Και θέλω να κάνω και ένα ερώτημα. Ε, κατά τη δική σας άποψη, αν ε, ας πούμε πάρετε τη Γενική Διεύθυνση και κάνετε εκεί κάποια σύγκριση με βάση τα δικά σας κριτήρια, ποια είναι η βέλτιστη πρακτική, τι θα συστήνατε στους μηχανισμούς ελέγχου, ε, στα λογιστικά, σε ποιους τομείς υπάρχει αυτό το βέλτιστο πρότυπο, ε, σε ποιους ακριβώς τομείς μπορούν να μάθουν άλλες γενικές διευθύνσεις, ας πούμε, από τη δική σας. Άλλα θέματα. Πάμε στην Όλαφ υπηρεσία καταπολέμησης απατών. Είχαμε μία συνέντευξη με τον Γενικό Διευθυντή της Όλαφ, τον κύριο Κέσλα, και μας ανέφερε ότι οι εγκληματίες επιλέγουν και στοχεύουν σε κράτη με τρωτή νομοθεσία απέναντι σε απάτες. Ας πούμε, Τσεχία, Ουγγαρία, εκείνος τα είπε, Ρουμανία, Ουγγαρία, αυτές έχουν τρωτή ε, νομοθεσία σε σχέση με τις απάτες. Εσείς τα ξέρετε αυτά. Τα ξέρετε αυτά που είπε ο Γενικός Διευθυντής της Όλαφ. Και αν τα ξέρετε, τι ακριβώς κάνετε για να τα αντιμετωπίσετε. Και τέλος και ένα άλλο ερώτημα που και αυτό αφορά την ε, Όλαφ για το θέμα Νταλή, του κυρίου Νταλή, του Επιτρόπου. Εδώ λοιπόν εσείς ως Επιτροπή ε, έχετε λάβει στα χέρια σας αρκετό υλικό και από το υλικό αυτό έχει προκύψει ότι υπάρχουν κάποια προβλήματα με την απαλλαγή του Επιτρόπου. Εμείς λοιπόν ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, δυστυχώς ε, δεν κληθήκαμε να τοποθετηθούμε και θέλω να σας πω δεν πιστεύετε εντάξει δεν λέω σε όλο το κοινοβούλιο, αλλά εν πάση δεν πιστεύετε ότι στο κοινοβούλιο υπάρχουν ε, άνθρωποι εχέμηθοι που θα μπορούσατε να τους συμπεριλάβετε σε τέτοιου είδους πληροφόρηση. Γιατί αλλιώ τι γίνεται. Απλά εμεί καλούμεθα να καταπίνουμε ορισμένα πράγματα, αλλά δεν είναι έτσι. Εμείς θα θέλαμε να ξέρουμε περισσότερα πράγματα, καλύτερη ενημέρωση, να είμαστε σίγουροι ότι σε τελική ανάλυση όλα αυτά που έγιναν και λέγονται για τον Επίτροπο είναι πράγματι τεκμηριωμένα. Το τελευταίο ερώτημα που θέλω να κάνω αφορά τα έγγραφα που σας είχαμε ζητήσει σχετικά με τη συμφωνία για τον καπνό. Μας απαντήσατε λοιπόν και μας είπατε ότι παρακαλώ διευκρινίστε την ερώτησή σας. Και εμείς τη διευκρινίσαμε. Μετά όμως εσείς μας δώσατε 24 έγγραφα και 16 περίπου σημειώσεις. Εντάξει, αυτά μπορεί κανείς να διαβάσει και διερωτώ γιατί μας είπατε να διευκρινίσουμε, αφού έτσι και αλλιώς κι εσείς μας δώσατε πολύ λιγά έγγραφα και λέτε αυτά είναι όλα και όλα αυτά που έχετε. Μήπως όμως υπάρχουν κι άλλα που δεν μας τα δώσατε. Θα ήθελα παρακαλώ να μας απαντήσετε από αυτού. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Πίπα. Ο κύριος Μούλντα έχει το λόγο. Uh, ευχαριστώ Πρόεδρε. Ενδιαφέρουσα συζήτηση. και εδώ έχω ήδη τις παρατηρήσεις του Επιτρόπου μετά τη συζήτηση. Μου τις έδωσαν ε, νωρίτερα, ε, χρήσιμο μεν. Θα ήθελα όμως να θέσω κάποιες ερωτήσεις και να κάνω κάποια σχόλια. Αρχικά, αναπόφευκτα, σήμερα αυτά που ασχολήσαμε, αποφασίσαμε τον Μάη περί απαλλαγής, μας ρώτησαν εφόσον παρέχουμε απαλλαγή, πώς μπορείτε να και το πράτεται διότι ακόμα και μετά από 18 χρόνια δεν κατέστη δυνατόν για την Κομισιόν να επιβεβαιώσει το λεκτικό συνέδριο και νομίζω ότι έχει φτάσει ο καιρός να αρνηθούμε την απαλλαγή διότι όπως θα θυμίστε η απαλλαγή όταν δεν χορηγήθηκε στο παρελθόν στην Κομισιόν χρειάστηκε να παρτιθεί και αυτό ήταν ένα καταστροφικό αποτέλεσμα. Εάν δείτε τα ψηφίσματα σχετικά με την απαλλαγή που ψήφισε το Κοινοβούλιο μας, μπορείτε να πείτε ότι υπάρχει ένα σταθερός παράγον από το 2003 και αυτό είναι το ότι το Κοινοβούλιο εντοπίζει ότι το πρόβλημα έγκυται στα κράτη-μέλη και πως τα κράτη-μέλη δεν επιθυμούν να συνεργαστούν επαρκώς με την Κομισιόν. Και θεωρώ πως οι παρατηρήσεις του συγητή περί αυτού είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες. Εκ πρώτης ματιάς προτίθεμαι να τις στηρίξω. Πολύ καλές λοιπόν οι προτάσεις του. Το Κοινοβούλιο εντόπισε ότι θα πρέπει να αναζητηθούν πολιτικές ευθύνες στα κράτη-μέλη και πως κάποιος θα πρέπει στο τέλος του οικονομικού έτους να θεωρηθεί υπεύθυνο για τα τεκτενόμενα. Και αν αυτό το πολιτικά υπεύθυνο άτομο κατά την άποψή του θεωρήσει ότι τα χρήματα σωστά δαπανήθηκαν Αυτό δεν ε, θα ήταν και πολύ καλό για την πολιτική του υγεία. Αυτό θεώρησε το Κοινοβούλιο λοιπόν σε ένα το 2006 όταν με το Συμβούλιο αποφασίσαμε πως αιτήσιες ε, συνόψεις θα υποβάλλονται και οι αιτήσεις αυτές τις συνόψεις ακολουθούσαν τις δηλώσεις των κρατών μελών ως ε, δήλωση του κράτου μέλους γιατί με το πώ δαπανέθηκαν τα χρήματα. Τώρα, η Κομισιόν μετά από όλα αυτά για το Συμβούλιο αποφάσισαν ότι αυτές οι συνόψεις ε, θα πρέπει να υποβάλλονται αλλά το Κοινοβούλιο δεν έχει καμία σχέση να αναμειχθεί με αυτές. Τώρα αυτές οι συνόψεις φυσικά έγιναν διαθέσιμες ε, στα μέλη της Επιτροπής μας και όταν μετέβην για να αναζητήσω αυτές τις συνόψεις ε, μάλιστα μου αφαιρέθηκε και το κινητό μου τηλέφωνο και διαπίστωσα ότι οι δηλώσεις αυτές, οι συνόψεις αυτές ήταν στην γλώσσα της ε, κάθε χώρας. Δηλαδή τα ελληνικά ήταν στα ελληνικά, τα αγγλικά στα αγγλικά και ούτω καθεξής. Πώς το καλό λοιπόν η Κομισιόν και τα κράτη-μέλη μπορούν να ισχυρίζονται πως ε, οι προθέσεις της ε, διαθεσμικής συμφωνίας πληρώθηκαν με την υποβολή αυτών των ε, συνόψεων. Γιατί όμως χρειάστηκε τόσος χρόνος που κατά την άποψή μου το αποτέλεσμα δεν ήταν και ιδιαίτερα επικοδομητικό. Έχουμε τώρα τον νέο δημοσιονομικό κανονισμό και αναφέρεται ο εθελοντικός χαρακτήρας αυτών των ε, δηλώσεων. Είναι εθελοντικός. Η Κομισιόν λοιπόν όμως θα πρέπει να εφαρμόσει. Διότι η αρμόδια τον προβλησμό αρχή θεωρεί ότι τα κράτη-μέλη χρειάζεται να λάβουν περαιτέρω ευθύνε. Και η Κομισιόν τη φορά αυτή δεν μπορεί να το αγνοήσει, όπω συνέβη με τι συνόψει αυτέ. Και ρωτώ, τι προτίθεται η Κομισιόν να πράξει ώστε να καταστεί πιο ελκυστικό για τα κράτη-μέλη να εκδίδουν αυτές τις ε, αιτήσει δηλώσεις. Έχουμε το παράδειγμα τριών κρατών. Η πρώτη ήταν οι κατοχώρες, ακολούθησε το Βασίλειο και η Σουηδία. Τι λοιπόν περί αυτού η Κομισιόν και κατά πόσον επιθυμεί να ενθαρρύνει και τα υπόλοιπα κρατημέλη και να πει ότι εμείς απαιτούμε από τα κράτη-μέλη η δήλωση να περιέχει το παρακάτω στοιχεία. Και ερώτησή μου ποιος ε, είναι αυτό ο χαρακτήρας των δηλώσεων και ποιο είναι το αποτέλεσμα, δηλαδή λιγότεροι έλεγχοι θα ασκούνται. Θα ήθελα λοιπόν μια σαφή απάντηση από την Κομισιόν τι προτείνεται να πράξει με αυτό το άρθρο στο νέο δημοσιονομικό κανονισμό που καθιστά εφικτό τα κράτη-μέλη να υποβάλουν αυτήν την δήλωση σε συνεργασία με τα εθνικά ελεκτικά συνέδρια. Αυτή νομίζω είναι η θέση του Κοινοβουλίου από το 2003. Τι προτίθεται λοιπόν να κάνει η Κομισιόν και μια παρατήρηση ως πολιτικοί θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί για το τι δηλώνουμε στα μέσα ενημέρωσης ε, δημοσιογράφους ε, των κατοχωρών αναφορικά με τις δαπάνες. Ε, δεν υπήρξαν κάποιες δηλώσεις που είχαν αρνητικό αντίκτυπο. θα έχουμε όμως κάποια παραδείγματα και ένα από αυτά τα παραδείγματα είναι ότι στην Πολωνία για τους αυτοκινητοδρόμους οι οποίοι κατασκευάστηκαν με κοινωτικά κονδύλια έχουν υποθετηθεί για κάποιες οθόνες και βλέπουμε ότι από τη μία πλευρά στην οθόνη παρουσιαζόταν ο αυτοκινητόδρομος Ακούγαμε ήχους και γιατί έχουμε αυτούς τους, τους ήχους που περιέχαν κάποιες φωνές και τι θα μπορούσε να μας απαντήσει γι' αυτό. Ο κύριος ε, Σκυλακάκης και μετά θα ακολουθήσουν και άλλοι ομιλητές. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ Επίτροπε. Επειδή οι συνάδελφοι και ο εισηγητή αλλά και οι συνάδελφοι που μίλησαν μετά από εκείνον ε, κάλυψαν ε, πολλά σημεία, ε, θα, κάνω, θα υποβάλω μόνο ένα ερώτημα επανερχόμενο σε ένα θέμα το οποίο με απασχολεί ιδιαίτερα Είπατε, Επίτροπε Σιμέτα, ότι κάνει να αναθεώρηση του ελεγκτικού περιβάλλοντος του για καλύτερη εστίαση στην περίπτωση απατών και στη μείωση των κινδύνων ο, το βασικό μας, ο βασικός μας τρόπος να, να αντιμετωπίσουμε την απάτη είναι η Όλαφ. Και σας είχα ρωτήσει όταν είχατε έρθει το Δεκέμβριο κατά πόσο μπορούμε να αυξήσουμε τις έρευνες ιδίας πρωτοβουλίας ε, για την Όλαφ και η απάντησή σας τότε ήταν θετική. Όμως επειδή μαθαίνω πράγματα, επαναλαμβάνω εγγράφω στην ερώτησή μου, επανάλαβα την ερώτησή μου και μετά η απάντησή σας ε, ήταν ε, αρνητική. Το ερώτημά μου είναι λοιπόν πάρα πολύ απλό, μία ακόμη φορά. Είδαμε ότι ένα τμήμα του ποσοστού σφάλματος, και αυτό είναι βέβαια μια θετική εξέλιξη, προέρχεται από ε, απάτες. Ε, υπάρχουν χώρες από τις οποίες, στις οποίες δεν υπάρχει κανένα τμήμα του ποσοστου σφαλματος και αυτο ειναι βεβαια μια θετικη εξελιξη προερχεται απο απατες ε σφάλματος που να έρχεται από την απάτη, που να προέρχεται από την απάτη. Και υπάρχουν χώρες ε, στις οποίες ε, γνωρίζουμε ότι τα πράγματα είναι διαφορετικά. Και ξέρουμε ότι αποτυγχάνουμε και δεν λέω ότι αυτό ισχύει μόνο σε μία χώρα, αλλά σε πολλές χώρες. Όμως, αυτή τη στιγμή δεν εστιάζουμε στον πραγματικό κίνδυνο, αλλά μόνο εκεί που μας ε, ενημερώνει, που μας λέει κάποιος ότι κάτι δεν πάει καλά. Και όταν κάποιος δεν μας λέει ότι κάτι δεν πάει καλά, η Όλαφ δεν ερευνά, δεν είναι παρούσα, ακόμα και αν υπάρχουν άλλα αποδεικτικά στοιχεία ε, που ε, υποδηλώνουν μεγάλο κίνδυνο. Πώς μπορεί λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λέει ότι θα παραμείνει μόνο σε αυτή την πολιτική ε, whistleblowing, ε, του να μας λέει δηλαδή κάποιος ότι ε, κάτι δεν πάει καλά, όταν υπάρχει κίνδυνο σε τόσους πολλούς τομείς. Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ λέει ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι ιδιαίτερα από εδώ και δύο χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνει ιδιαίτερη προσοχή όχι μόνο στην νομιμότητα των ε, δαπανών αλλά και στις επιδόσεις. Επίσης ε, είμαι ευγνώμων και στο ελεγκτικό συνέδριο γιατί πραγματικά το, παρακολουθούν ε, πολύ σοβαρά. Βλέπουμε ότι υπάρχουν βελτιώσεις ε, από την πρώτη χρονιά που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε ιδιαίτερη προσοχή στις επιδόσεις, όμως σύμφωνα με το ελεγκτικό συνέδριο και πάλι δεν είναι αυτό το οποίο θα μπορούσαμε να περιμένουμε ακόμα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και το ερώτημά μου έχει να κάνει ακριβώς με αυτό. Φοβούμαι και θα ήθελα να πω ότι μάλλον αυτό σχετίζεται με αυτά που είπε ο συνάδελφος Μούλντερ για, τα, για την ηχομόνωση στους αυτοκινητοδρόμους στην Πολωνία. Το γεγονός δηλαδή ότι πολλά χρήματα ξοδεύονται σε μερικές χώρες με έναν τρόπο που πιστεύουμε ότι τέλος πάντων, άμα το πω έτσι με έντονους όρους, γελίο και τέλος πάντων με υπιότερους ε, όρους ε, δεν είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικός, τέλος πάντων δεν εξυπηρετεί τον οικονομικό στόχο που θα περίμενε κανείς, το ερώτημά μου δεν αφορά άμεσα το ρόλο της Επιτροπής, αλλά το ρόλο των κρατών μελών περισσότερο και το βλέπουμε αυτό σε όλε τι ειδικέ εκθέσει του ελεγκτικού συνεδρίου. Το είδαμε την περασμένη εβδομάδα σε μια ειδική έκθεση για ε, τις δαπάνες για την ενεργειακή αποτελεσματικότητα που φαίνεται ότι δεν ενδιαφέρονται οι χώρε για την ενεργειακή αποδοτικότητα, ενδιαφέρονται για τα ευρώ που ξοδεύονται στη δική του χώρα. Βάσει αυτών των εκθέσεων, λοιπόν, χρηματοδοτούνται προγράμματα με ευρωπαϊκά κονδύλια υπό την ευθύνη των κρατών μελών όμως με επιστροφή στην επένδυση 150 χρόνων περίπου, που κάτι το οποίο μου φαίνεται μάλλον γελίο. Το ερώτημά μου λοιπόν έχει να κάνει πολύ περισσότερο με την ελευθερία, την ευελιξία που επιτρέπουμε στα κράτη-μέλη ε, κατά την ε, αξιοποίηση των κονδυλίων. Εγώ είμαι υπέρ των ευρωπαϊκών ε, ε, κονδυλίων, αλλά είναι κάτι που προφανώς δεν μπορούμε να τα αφήσουμε μόνο στα χέρια των κρατών μελών ε, χωρίς μεγαλύτερη επιτήρηση από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εγώ σε σχέση με το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο ε, θα ε, στεναχωριόμουν πραγματικά να βλέπουμε πολύ μεγαλύτερη επιλεξιμότητα μεταξύ των κονδυλίων που ξοδεύονται και της αποτελεσματικότητας ε, των προγραμμάτων. Θα με στεναχωρούσε αν δεν συνέβαινε κάτι τέτοιο. Και δεδομένων των παραδειγμάτων που έχουμε και δεδομένου του γεγονότος ότι πολύ περισσότερη σημασία δίνει πλέον η Επιτροπή στις επιδόσεις, είστε διτεθειμένος να δώσετε μία ακόμη όθηση σε αυτό το θέμα, να γίνεται, μία, να γίνεται σοβαρός έλεγχος, να γίνεται μία σοβαρή εξέταση των επιδόσεων και της ε, αποτελεσματικότητας των δαπανών, είστε διατεθειμένος να παρέμβετε ακόμη και σε αυτό το τελευταίο τελικό στάδιο διαπραγματεύσεων ε, για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, να παρέμβετε πολύ πιο ε, σοβαρά σε σχέση με το θέμα αυτό της επιλεξιμότητας ε, γιατί επειδή εγώ έρχομαι από μάλλον ε, το πιο το κόμμα της Ολλανδίας που είναι, υπέρ, το, που είναι περισσότερο υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να πω ότι βλέπουμε ακόμη κάποια παραδείγματα πολύ κακής αξιοποίησης των κονδυλίων. Ο κύριος Στάς. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να συμφωνήσω σε σχέση με την ε, σημασία του ρόλου των κρατών μελών και των προσπαθειών που καταβάλουμε τα τελευταία χρόνια να ε, έχουν μεγαλύτερη ευθύνη τα κράτη-μέλη. Άκουσα τα λεγόμενα του ελεγκτικού συνεδρίου Μπορούμε να έχουμε προγράμματα από το 2000 ως τώρα και με βάση έκθεση του συνεδρίου να προκύπτει ότι οι προθεσμίες ε, για τις επενδύσεις να ε, καθυστερούν τόσο πολύ. Δηλαδή, μίλησε ο κύριος Γερμπράντ για αυτό το θέμα λέγοντας ότι κάποια ε, προγράμματα μπορεί να αποδώσουν καρπούς 150 χρόνια. Υπάρχουν και χειρότερα παραδείγματα. Είπατε βέβαια ότι οι αξιολογήσεις είναι πολύ σημαντικές και ότι πρέπει να δούμε την προστιθέμενη αξία αν δεν υπάρχει μία, ε, ούτε μια υπηρεσία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή που να μπορεί να το παρακολουθεί αυτό, δεν έχει νόημα. Ε, πρέπει να γίνεται μια εσωτερική αξιολόγηση αυτών των προγραμμάτων. Μήπως θα ήταν χρήσιμο αυτές οι εκθέσεις ε, να είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο, ώστε να είναι κάπως πιο διαφανείς. Και συνεπώς οι συνάδελφοι ή ομάδες δράσης που θέλουν να εξασφαλίσουν ότι βαπανώνται σωστά τα χρήματα αυτά, να ε, μπορούν ε, να ε, είναι κάποιο είδους φύλακες, να βρουν ως φύλακες κατά κάποιο τρόπο. Από τις εκθέσεις αυτές μαθαίνουμε πολλά πράγματα. Εμείς ως Επιτροπή ασχολούμαστε, ασχολούμαστε περισσότερο με τις εκθέσεις του ελεγκτικού συνεδρίου και αναρωτιόμαστε πώς μπορούμε να τις αξιοποιήσουμε καλύτερα. Αναρωτιέμαι όμως αυτές οι ειδικέ εκθέσεις τι ε, συνέχεια λαμβάνουν ε, αν υπάρχει μια ειδική έκθεση, για παράδειγμα, για την εξοικονόμηση ενέργειας. Αυτό στη συνέχεια ε, φτάνει μέχρι τον Επίτροπο, τον Υπεύθυνο για την Ενέργεια ή εσείς είστε εκείνος που θα ασχοληθεί πρώτα με το θέμα αυτό. Και ένα ερώτημα ακόμη. Χρόνια επεξεργαζόμαστε την απαλλαγή για το Συμβούλιο και το Συμβούλιο θεωρεί ότι ο προϋπολογισμός του είναι τμήμα ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ότι δεν χρειάζεται να μας διαθέτουν τα σχετικά στοιχεία και ότι δεν χρειάζεται να δώσουμε απαλλαγή για τον προϋπολογισμό του Συμβουλίου. Εσείς συμφωνείτε με αυτή την ερμηνεία ε, που κάνει το Συμβούλιο και αν συμφωνείτε με αυτή την ερμηνεία πρέπει να σας ε, ρωτήσω ως εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Επιτροπής εσείς θα μπορούσατε να πάτε στο Συμβούλιο και να πείτε θα ήθελα αυτό και εκείνο το έγγραφο που έχει να κάνει με τον προεπολογισμό του Συμβουλίου. Γιατί δεν μπορεί να υπάρξει απαλλαγή παρά μόνο αν έχουμε στη διάθεσή μας αυτά τα έγγραφα. Ή αν δεν συμφωνείτε με αυτήν την ερμηνεία του Συμβουλίου, πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε να επιλύσουμε το πρόβλημα αυτό. Και κάτι ακόμη, το οποίο συνδέεται με το θέμα του κυρίου Πίπερ, για τις, ε, τις έρευνες της Όλαφ, ε, για τον ε, πρώην επίτροπο Ντάλι και, τον, και, του, και τους φίλους του, που ήθελε να λάβει χρήματα για να επηρεάσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είστε υπεύθυνο και για την όλα σε τελική ανάλυση και συμφωνείτε με την ερμηνεία αυτή ε, της νομικής υπηρεσίας του Κοινοβουλίου βάσει της οποίας εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να έχουμε πρόσβαση στις σχετικές έρευνες της Όλαφ. Μη μας πείτε ότι ναι, αλλά γίνεται και έρευνα στη Μάλτα, οπότε δεν χρειάζεται. Ένα από τα πλεονεκτήματα του να είναι κανεί ε, στο Κοινοβούλιο και σε αυτή την Επιτροπή ε, πολλά χρόνια είναι ότι έχει ζήσει κανεί ε, πολλά σκάνδαλα. Ο κύριο Μόλντερ και εγώ είμαστε πολλά χρόνια εδώ. Θα θυμάστε το 2003 μία υπόθεση Eurostat, υπήρχαν έρευνες στη Γαλλία στο Λουξεμβούργο και παρόλα αυτά ο Επίτροπος Πρόντι τότε είχε διαθέσει τα σχετικά έγγραφα στο Κοινοβούλιο. Υπάρχει λοιπόν ένα προηγούμενο μία δικαστική έρευνα και παρόλα αυτά εμείς είχαμε πρόσβαση στα έγγραφα. Για ποιο λόγο λοιπόν εμείς ως μέλη της Επιτροπής αυτής δεν μπορούμε να δούμε τα έγγραφα που αφορούν την υπόθεση Ντάλι. Της 11 Δεκεμβρίου αποστήλαμε ε, μια επιστολή στην οποία λέγαμε ότι μπορεί να υπάρχουν κάποια προβλήματα με την έρευνα τη Όλαφ ενδεχόμενα προβλήματα. Τι σημαίνει δηλαδή ότι δεν ακολουθήθηκαν κάποιοι κανόνες, ότι υπήρχαν άλλε παρατυπίες. Τι σημαίνει ακριβώς. Μήπως ε, δεν ήταν απόρριτη τελικά η έρευνα. Ποιο ακριβώ ήταν το πρόβλημα. Εσείς είστε υπεύθυνος για αυτό το θέμα. Και τι μέσα έχετε στη διάθεσή σας να λάβετε δράση αν μια εποπτική επιτροπή σας ζητήσει κάτι τέτοιο, αν σας πει δηλαδή κάποιος ότι υπάρχουν προβλήματα με μια έρευνα. Θα ήθελα να μάθω λοιπόν αν ε, έγινε κάτι σχετικά με αυτό. Σας ζητήσαμε τεκμηρίωση, μας είπατε είναι πάρα πολύ η τεκμηρίωση, τελικά λάβαμε 24 έγγραφα. Σε σχέση με τον καπνό. Υπήρχε και μία ερώτηση, στις ερωτήσεις που σας υποβάλαμε, ο κύριος Πετίτ που είναι μάλιστα και πρόεδρος της Επιτροπής Διοντολογίας ε, και εξετάζει όλα αυτά τα έγγραφα. Τρεις ε, προϋποθέσεις υπήρχαν, ε, εμπειρογνωμοσύνη, γνώση του θέματος και αμεροληψία. Πώς μπορείτε να πείτε ότι ο κύριος Πετή είναι αμερόληπτος, είναι δικηγόρος πολλών καπνοπαραγωγών. Πώς είναι λοιπόν δυνατόν ένας τέτοιος άνθρωπος, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πολύ εξοικειωμένος δεν λέω, γνωρίζει το θέμα. Αλλά πώς μπορείτε να πείτε ότι ένας άνθρωπος που είναι σε αυτή τη θέση είναι πραγματικά μερόληπτος. Αυτή είναι η τελευταία μου ερώτηση. Ευχαριστούμε πολύ. Κυρία Αντρεάσεν. Thank you, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όπως και ο Πίπερς, Πίπερς να πω και εγώ, πως ως συνήθως, η ε, την τελευταία δεκαετία τουλάχιστον, η Επιτροπή επικρίνει τα, τα κράτη-μέλη για τις παρατυπίες τους. Θα ήθελα να λάβω μια συγκεκριμένη απάντηση από σας Δηλαδή για ποιο λόγο η Κομισιόν δεν μπορεί να εγκρίνει τους ε, κανόνες επιλεξιμότητας που έχουν θέσει τα κράτη-μέλη. Γιατί η Κομισιόν θέλει να τους αναθεωρήσει και να παρεμβαίνει αν κρίνει ότι αυτοί οι κανόνες επιλεξιμότητας δεν είναι αποτελεσματικοί ή δεν επιτρέπουν την κατάλληλη τη σωστή χρήση των πόρων. Γιατί η Κομισιόν επίσης πρέπει να αναλάβει κάποιες πρωτοβουλίε για την απλούστευση αυτών των κανόνων. Φαίνεται όμω πω η διαδικασία, νόμιζα ότι η διαδικασία είχε ολοκληρωθεί. Αλλά φαίνεται ότι δεν έχουν έτσι τα πράγματα. Τώρα, σε σχέση με την ανάκτηση, να πω πως ε, οι ανακτήσεις δεν αντικαθιστούν τους ελέγχους, αποτελεσματικούς ελέγχους. Το γεγονό ότι ανακτούμε τα χρήματα, αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί να είμαστε ικανοποιημένοι από τους ελέγχους που ασκούμε. Μπορούμε να ε, κάνουμε τα μέτρα πιο αυστηρά και τους κανόνες αυστηρότερους αν θέλουμε να βελτιώσουμε τους, την ανάκτηση πόρων. Είπατε ότι το, 1900, το 2011 ε, ανακτήσαμε 1,84 δις. Μετά από πόσα χρόνια ανακτήσαμε αυτά τα κονδύλια. Δεν έχει νόημα να μας πείτε ότι ανακτήσαμε τεράστια ποσά και πως αυτό αντιπροσωπεύει κάτι παραπάνω από το 1% του ετήσιου προπολισμού για το 2011. Ίσως ε, να ε, αντιπροσωπεύει 5 ή 6 έτη παρατυπιών Θεωρώ ότι δεν είναι και τόσο υψηλό το ποσοστό ανάκτηση. Τώρα, μέσα σε ένα άλλο σημείο σε σχέση με τι ανακτήσει είναι ότι τι περισσότερε φορέ τα χρήματα δίνονται από τις εθνικές κυβερνήσεις, οι οποίες δεν είναι ιδιαίτερα επιτυχείς στην ανάκτηση κονδύλιων από τους διότι η Κομισιόν χορηγεί χρήματα σε κάποιους οργανισμούς και κατά ανάγκη αυτά τα χρήματα δεν πάνε στην κεντρική κυβέρνηση. και αν και τις κυβερνήσει δεν μπορούν να ανακτήσουν τα χρήματα αυτά από τους δικαιούχου, αυτό σημαίνει ότι ο φορολογούμενος πληρώνει δύο φορές το μάρμαρο. Τέλος, το τομέα της έρευνας. Πολλές κριτικές ακούγονται τα κρατημέλη σχετικά με την κοινή διαχείριση. Αλλά η διαχείριση αυτή γίνεται από την Κομισιόν στην ουσία. Λοιπόν, πώς είναι δυνατόν να έχουμε αυτό το ανεξάρτητο πιστοποιητικό των ελεκτικών αρχών, αλλά το ελεκτικό συνέδριο θεωρεί ότι το 80% έχουν επηρεαστεί από σοβαρά λάθη. Ευχαριστώ. Ο Ευχαριστώ, Πρόεδρε, ευχαριστώ, Επίτροπε, για τι επιπλέον πληροφορίε και προ το Ελεκτικό Συνέδριο. Ευχαριστώ για τι παρεμβάσεις του. Προσωπικά χαίρομαι με αυτή τη συζήτηση, διότι παρατηρούμε πω ε, μετά από την, με την περιπλοκότητα των κανόνων που υπάρχουν, με τι πολλαπλέ προσχωρήσει χωρών μελών τα τελευταία χρόνια. Το δημόσιο χρήμα το οποίο συνδέεται με απάτες και με καταχρήσεις αλλά και με διαφθορά όλα αυτά πραγματικά καταστούν τα θεσμικά όργανα λίγο νευρικά, διότι η κοινή γνώμη περιμένει απαντήσει. Και ειδικά τι κάνουμε τα τελευταία 5-6 χρόνια και δι η Επιτροπή Ελέγχου Προπολογισμών. Ε, τη ζήτηση αυτή την έχουμε ήδη κάνει και πρέπει να αναρωτηθούμε κατά πόσον δεν έχουμε ένα σύστημα το οποίο εκπνέει λίστια. Και αμφισβητούμε τώρα τα κράτη-μέλη. Αυτά τα δυστυχή κράτη-μέλη και τα υπουργεία τους ε, όλοι λένε θέλω τα χρήματά μου πίσω. Με τα ευρωπαϊκά χρήματα συχνά το δωτώ κάποιες ε, περιφερειακές ε, δραστηριότητες κλπ. αλλά και εθνικές. Νομίζω ότι έφτασε η στιγμή όπου η Ευρώπη θα πρέπει να ανακτήσει τα χρήματά της. Δεν πιστεύω σε αυτήν την ιστορία των ε, δηλώσεων αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων συχνά το δήλωσα σχέση προς τους συναδέλφους μου και έτσι και το υποθέσουμε ότι το πράττουν αυτό και σε ό,τι αφορά όμως τα αποδεικτικά στοιχεία κατά τον έλεγχο δεν ε, είναι αποτελεσματικά όταν του ζητούμε να μας ε, να συνεργαστούν με τις διοικήσεις τους, τα υπουργεία τους και ε, να θέτουν όλες τις δυνατότητε τους στο ελεκτικό συνέδριο και να κάνουν μια δήλωση. Εγώ δεν βλέπω να υπάρχει κάποιο νόημα, αλλά να πρέπει να συμπεριληφθούν τα εθνικά ελεκτικά συνέδρια στον έλεγχο. Διότι αυτά είναι ανεξάρτητα σχέση με τους υπουργούς και, τους, και τις κυβερνήσεις. Εδώ θα έχουμε κάποιο ενδιαφέρον. Τώρα, άρνηση απαλλαγή, γιατί όχι, αρνηθήκαμε την απαλλαγή στο παρελθόν. Τι έγινε, τίποτα. Το Συμβούλιο παρετήθηκε, το Συμβούλιο παίρνει το λόγο, ενδιαφέρεται. Θα έχουμε συζητήσει την Ολομέλεια και δεν θα είναι καν παρόν. Το Συμβούλιο δεν εκπροσωπεί τα κράτη-μέλη, δεν είναι μια οντότητα που εκπροσωπεί τα κράτη-μέλη, αλλά στο Συμβούλιο έχουμε τους υπουργούς που ε, διευθύνουν και δίνουν εντολές στις διοικήσεις ε, και μετά κάνουν τα ασφάλματα τα οποία όλοι γνωρίζουμε και τα οποία λυπούμεθα. Και θα είχαμε κάθε συμφέρον να έχουμε μια συζήτηση για αυτή την διαδικασία απαλλαγή με το ελεγκτικό συνέδριο, το ευρωπαϊκό φυσικά, αλλά το, το ελεγκτικό συνέδριο μας λέει ότι έχουμε μία δήλωση διαβεβαίωσης, διασφάλισης, αλλά έχουμε και τέσσερις ε, γνωμοδοτήσεις ε, των ε, ελεγκτών για έναν βουλευτή, ειλικρινά τώρα. Ε, για Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή για την Επιτροπή μας να πούμε ότι έχουμε μια θετική ή αρνητική δήλωση είναι αδύνατον. Έχουμε τέσσερις γνωμοδοτήσεις και θα θέλαμε αυτή η δήλωση διασφάλισης ε, αν είναι θετική ή έχει κάποιες επιφυλάξεις και μετά θα μπορούσαμε να πούμε αν αυτή η δήλωση είναι αρνητική τότε το αποτέλεσμα θα είναι να διώξουμε την Κομισιόν και να ψηφίσουμε μια πρόταση μορφής. Εξάλλου, ανά πάση στιγμή μπορούμε να ε, ε, κάνουμε πρόταση μορφή προ την Κομισιόν, αλλά δεν είναι απαραίτητο κατά την άποψή μου, αλλά το σύστημα δεν είναι σωστό, δεν είναι ορθό. Δεν αναλύονται επαρκώ οι αδυναμίε ενό συστήματο που κατά την άποψή μου είναι τα ταλίστια, επαναλαμβάνω. Ε, και τώρα επαναλαμβάνω την ε, αρχική μου θέση να έχουμε μια μεγάλη συζήτηση με το ελεκτικό συνέδριο, τους εκπροσώπους των εθνικών ελεκτικών συνεδρίων, τα εθνικά κοινοβούλια που θα πρέπει να ελέγχουν τις κυβερνήσεις τους, την Επιτροπή μας, ε, τις ελεκτικές αρχές και από κοινού να εξετάσουμε την λειτουργία των ευρωπαϊκών ε, οικονομικών, ε, των ευρωπαϊκών δημοσιονομικών, να πάμε βρούμε ένα σύστημα λίγο πιο απλό και να επανακτήσουμε τις διαδικασίες χρηματοδότησης ε, με ελέγχους πόσο κοστίζει αυτή η διαχείριση, είναι αποτελεσματικά ή όχι, αν δεν είναι, να την καταργήσουμε είχαμε μια συζήτηση με τον κύριο Άστον, που είναι και αντιπρόεδρο τη Επιτροπή. Και είχαμε πει θα δώσουμε την απαλλαγή στην υπηρεσία εξωτερική ε, <clears throat> δράση. Πάνω σε τι θα, θα βασιστούμε, σε, στα διοικητικά θέματα ή και τα λειτουργικά έξοδα. Πρέπει να το ε, εξηγήσουμε αυτό, διότι υπάρχει παρα, παρεξήγηση με το Συμβούλιο, θα έχουμε και παρεξήγηση και παρανόηση με την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, διότι εδώ υπάρχουν δράσεις διακρατικές, ε, ποιες δώσει την απαλλαγή. Ε, Τα Εθνικά Κοινοβούλια, το Ευρωκοινοβούλιο και τι θα γίνει και αυτοί που θα κερδίσουν θα είναι οι αντιευρωπαίοι που θα πούνε να κοιτάξτε το σύστημα δεν λειτουργεί. Λοιπόν, εγώ προτείνω να προβληματιστούμε από κοινού και να αναθεωρήσουμε το σύστημα που είπα Ιταλία Ιταλίστη. ευχαριστώ. Ε, βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει ένα μεγάλο φάσμα μιλητών από τον κύριο Γκάιερ μέχρι τους συναδέλφους που έκαναν όλες αυτές τις ερωτήσεις. Και συνοψίζοντας, εγώ θα ήθελα να πω το εξής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μερικές φορές ε, αντιμετωπίζει το πρόβλημα ότι εδώ υπάρχει δημοκρατικό έλλειμμα δεν πρέπει να δίδονται χρήματα φορολογουμένων χωρίς ε, δημόσιο έλεγχο. Και όταν ε, το ελεγκτικό συνέδριο κάνει παρατηρήσεις. Είναι προφανές ότι πρέπει να ασχοληθούμε εμείς με όλα αυτά και δεν χρειάζεται να δικαιολογούμεθα αγαπητοί συνάδελφοι. Όταν δημόσια αναφέρεται ότι υπάρχει έλλειψη δημοκρατικού, ότι υπάρχει δημοκρατικό έλλειμμα, αυτό ε, δεν μπορεί κανείς να το απευθύνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και σίγουρα όχι σε εμά. Γιατί εμείς είμαστε εκείνοι που διεξάγουμε τους ελέγχους. Και εδώ ένα δεύτερο ερώτημα, το οποίο το έθιξαν αρκετοί συνάδελφοι σε σχέση με το αίτημα ενημέρωσης ε, στο πλαίσιο της διοργανικής συμφωνίας που έχουμε συνάψει με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όλα αυτά σε σχέση πάλι με την έκθεση της ε, Όλαφ για την παρέτηση του κυρίου Ντάλι. Μας λένε λοιπόν ότι πρέπει να δείχνουμε εμπιστοσύνη, ότι όλα έγιναν όπως προβλέπεται από τον νόμο, αλλά ε, τι σημαίνει αυτό. Ε, εντάξει, υπάρχει μια συμφωνία, μια διοργανική συμφωνία και όπως είπαν και πολλοί συνάλφοι και στον Φρανσου Πικ ε, και εκεί ε, την είδαμε την έκθεση ε, που είχε συσταθεί. Όσο περισσότερο καιρό δεν μας δείχνεται την έκθεση αυτή, τόσο περισσότερο και οι συνάδελφοι υποψιάζονται ότι κάτι δεν πάει καλά. Εγώ λοιπόν πιστεύω ότι αν όλα έγιναν όπως προβλέπονται, σίγουρα δεν θα υπήρξε πρόβλημα, αλλά φαντάζομαι ότι υπάρχει και μια διαδικασία που προβλέπει πως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα του, γιατί εμείς είμαστε ο θεσμός εκείνος που εκλέγεται άμεσα από, το, από τους πολίτες. Και κάτι άλλο, το τελευταίο που έχει σχέση με την απαλλαγή του Συμβουλίου. Εμείς ε, καλούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διαδραματίσει σημαντικότερο ρόλο, γιατί ξέρετε τι γίνεται, το ε, Συμβουλίο μας παραπέμπει στην Κομισιόν και λέει αφού απαλλάσσει την Κομισιόν δεν χρειάζεται έξτρα απαλλαγή του Συμβουλίου. Αυτό μας δεν είναι σωστό γιατί εμείς ε, μέχρι τώρα ε, δεν θέλαμε να μπλέξουμε την Κομισιόν στην απαλλαγή του Συμβουλίου. Και σε τελική ανάλυση ίσως το μόνο που μας απομένει είναι την ε, απαλλαγή του Συμβουλίου να την παραπέμψουμε και εμείς στην Κομισιόν. Θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει να ε, σταλεί ένα μήνυμα προς το Συμβούλιο ότι πρέπει να βρούμε κάποια λύση. Νομίζω λοιπόν ότι ομιλώ εξ ονόματος του συνόλου της Επιτροπής ότι ενδιαφερόμεθα για μια ουσιαστική λύση. Ευχαριστούμε πολύ ο κύριος Επίτροπος μέτα, ίσως ε, μπορεί να τοποθετηθεί στα θέματα που ετέθησαν. Ε, ίσως μπορείτε να δώσετε κάποιες απαντήσεις. Ευχαριστώ πολύ για όλα τα ερωτήματα. Πολλά ήταν βέβαια και κάλυψαν μεγάλη εμβέλεια θεμάτων, αλλά θα ήθελα να αρχίσω με κάποια σχόλια για όσα έθεσε ο κύριος Γκάιερ. Πρώτα απ' όλα το θέμα των εσόδων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποδίδει ιδιαίτερη προσοχή στη βελτίωση της κατάστασης στα τελωνία και προσπαθεί να εφαρμόσει μέτρα ε, διαφόρων ε, παραβιάσεων αντιμετώπιση διαφόρων παραβιάσεων. Αν δείτε και τα γραπτά μου, τη γραπτή μου απάντηση όσον αφορά τα τελωνία, ε, κάναμε πολύ σημαντική ε, προσπάθεια βελτίωσης της τελωνιακής διαδικασίας και τώρα παρακολουθούμε την εφαρμογή των μέτρων που έχουν ληφθεί προκειμένου να εξασφαλίσουμε ότι αυτή η απλοποιημένη διαδικασία δεν δημιουργεί περαιτέρω προβλήματα. Επίσης θέσατε το θέμα της καθυστέρησης του εξυγχρονισμού δεν είναι ακριβώς όμως ε, τα πράγματα ε, έτσι. Εμείς διαπραγματευόμαστε και με το Κοινοβούλιο και με το Συμβούλιο έναν ε, ενωσιακό τελωνιακό κώδικα που θα υποκαταστήσει τον εξυγχρονισμένο τελωνιακό κώδικα. Είναι γεγονός ότι ο προηγούμενος εξυγχρονισμένος τελωνιακός κώδικας προέβλεπε ε, εφαρμογή από τον Ιούνιο του 2013 του νέου κώδικα, αλλά λόγω της κρίσεως όλοι οι παράγοντες, ε, τα κρατημέλη, ε, οι έμποροι στους οποίους απευθυνόταν κατά κύριο λόγο αυτή η πρόταση, όπως επίσης και άλλοι εμπλεκόμενοι παράγοντες, πρότειναν να αναβάλουμε λίγο την ε, εφαρμογή του νέου κώδικα. Γι' αυτό ακριβώς προέκυψε η συγκεκριμένη πρόταση. Δεν είναι ακριβώς ε, σωστό ότι θα αρχίσει να ισχύει ε, το 2020. Ευθύς αμέσως θα αρχίσει να ισχύει μετά την έγκρισή του. θα αναπτυχθούν προοδευτικά τα αντίστοιχα ε, συστήματα πληροφορικής. Υπάρχει μάλιστα και ένας χάρτης πορείας ε, που έχει συμφωνήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τα κράτη-μέλη για το πότε και ποια συγκεκριμένη διαδικασία θα αρχίσει να ισχύει κατά το 2013 ε, και μετά το 2020. Αυτός ο κώδικας, ο τελωνιακός, είναι πάρα πολύ σημαντικός ε, και πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη και από το Κοινοβούλιο και από το Συμβούλιο σε ε, εύλογο χρονικό διάστημα πρέπει να εγκριθεί. Διαφορετικά θα δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στα τελωνία μετά από την 21η Ιουνίου του 2013. Ξέρετε ότι έχουμε μία νέα στρατηγική για το φόρο τη θέμενη αξίας και τώρα θα μπούμε στη διαδικασία υποβολής συγκεκριμένων προτάσεων. Πέρσι υποβάλαμε την πρόταση των ε, ε, της έγκαιρης ε, προειδοποίησης σε σχέση με τους, τις σχετικές παραβιάσεις ε, της απάτες στο φόρο προστιθέμενης αξίας. Τώρα προσπαθούμε να έχουμε ένα μηχανισμό αντιστροφής του άχθους της απόδειξης, κάτι το οποίο μπορεί να είναι πολύ σημαντικό για τις απάτες τύπου καρουσέλ και ε, νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό σε σχέση με την ανάπτυξη της δραστηριότητας της Eurofisk. Τώρα περνάμε σε αυτοματοποιημένη πρόσβαση σε πληροφορίες που αφορούν το ΦΠΑ, ε, από πλευράς κρατών μελών εννοώ. Όλα αυτά λοιπόν είναι μέτρα τα οποία βεβαίως είναι πάρα πολύ σημαντικά και είναι πάρα πολύ σημαντικό τα κράτη-μέλη να εγκρίνουν τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε σχέση, πούμε, με το μηχανισμό άμεσης αντίδρασης. Όλα τα κράτη-μέλη υποστήριξαν σε πολύ μεγάλο βαθμό την πρόταση επί της αρχής, αλλά όταν περάσαμε στην έγκριση, κάποια από αυτά τα κράτη-μέλη τουλάχιστον ε, φρονούσαν ότι κάτι θα έχαναν με την πρόταση αυτή και τελικά είμαστε τώρα ε, ακόμη στη διαδικασία διαπραγμάτευσης. Ε, αντί, λοιπόν να αντεγκρίνουμε τώρα την πρόταση ε, και να μπορέσουμε να ε, καταπολεμήσουμε επιτέλους την απάτη ΦΠΑ, ακόμα διαπραγματευόμαστε. Τώρα όσον αφορά τα φιλοσοφικά σας ερωτήματα, σε σχέση με την αντιμετώπιση των μεθοδολογικών ε, διαφορών μεταξύ του συνεδρίου, του Ελληνικού Συνεδρίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ναι, υπάρχουν κάποιες μεθοδολογικές διαφορές όντως και δεν ήθελα να σχολιάσω ειδικότερα τη μεθοδολογία του ελεγκτικού συνεδρίου πρέπει να την σεβαστούμε παρά το γεγονός, όπως είπατε, ότι το το θέμα τη 100% ποσοτικοποίηση των σφαλμάτων. Προφανώ είχατε στο μυαλό σα το θέμα των δημοσίων προμηθειών, όπου ακολουθήσαμε μια διαφορετική προσέγγιση. Αλλά τέλο πάντων δεν ε, ε αμφισβητούμε εμεί την ε, διαδικασία των, ε, που ακολούθησε το ελεγκτικό συνέδριο. Απλώ εμεί είχαμε μια προσέγγιση που αφορούσε περισσότερο τη ζημία που ε, προήλθε από την άτυπη χρήση των, ε, την παράτυπη χρήση των κονδυλίων για, τα, για τις δημόσιες προμήθειες ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι αν υπάρχει ε, παραβίαση αυτών των κανόνων αυτό είναι ένα θέμα που οδηγεί σε αυτό το 100% ποσοτικοποίηση που σας ανέφερα προηγουμένως αλλά σε σχέση με την συνολική προσέγγιση, την ευρύτερη προσέγγιση και τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να ε, προχωρήσουμε, πρέπει να συνεχίσουμε τη συζήτηση, ε, ενδεχομένως και όλας να την εμβαθύνουμε, σε σχέση με τον πολιετή χαρακτήρα των ελέγχων μας ε, και τη σημασία των υπολείπων λαθών, γίνεται τώρα πολύ τεράστια προσπάθεια προκειμένου να μπορέσουμε να εντοπίσουμε τι ανακτήσεις και τι διορθώσεις ε, πρέπει να ε, αποδοθούν σε ένα συγκεκριμένο έτος και αυτό απαντά και την ερώτηση της κυρίας Ανδρέασεν είναι γεγονός ότι μέχρι τώρα ήταν δύσκολο ε, να μην πω αδύνατο οι ανακτήσεις και οι διορθώσεις να αποδοθούν σε συγκεκριμένο έτος, όμως Από την επόμενη διαδικασία απαλλαγής, χορήγησης απαλλαγής, ε, ο υπεύθυνο λογιστικών ε, μας είπε ότι θα μας παρουσιάσει πληροφορίες ε, με την κατανομή ανάλογα με το έτος. Το σχόλιο μου όμως εδώ είναι το εξής, ότι το 2011 Όντως είχαμε ανακτήσει σε 1,84 δις το 2011. Δεν πρέπει να ξεχνάτε όμως ότι έγιναν και το 2009 και το 2010 και το 2008 και άλλα χρόνια έγιναν ανακτήσεις και διορθώσεις. Άρα δεν είναι κάτι το οποίο συμβαίνει άπαξ. Θέλουμε λοιπόν να βελτιώσουμε αυτές τις πληροφορίες και με τη βελτίωση αυτή Νομίζω ότι να δούμε πώς θα μπορούσαμε να συζητήσουμε μετά και αυτές οι πληροφορίες, πώς μπορούν να αντικατοπτρίζονται, να συμπεριλαμβάνονται και στη γνωμοδότηση του ελεγκτικού συνεδρίου. Υπήρχαν και κάποια άλλα ερωτήματα που αφορούσαν ε, την ε, επόμενη γενεά προγραμμάτων Κύριε Γκάιερ, θέσατε το θέμα των αναδρομικών προγραμμάτων, των καθαρών διορθώσεων. Ο κύριος Γκερμπράντε θέσε το θέμα της επιλεξιμότητας των προγραμμάτων. Όλα αυτά τα μέτρα παρουσιάζονται στα προγράμματα ναι, ε, της επόμενης γενεάς. Αυτή τη στιγμή είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο. Κάποιο μου ζήτησε να δώσω μεγαλύτερη όφηση. Είναι όμω πρόταση επιτροπή. Εμεί υποβάλαμε την πρόταση. Τώρα γίνονται οι διαπραγματεύσει μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου. Μεταξύ των ε, συνομοθετών. Και τώρα είναι στα δικά τους χέρια να αποφασίσουν ε, και να εγκρίνουν ε, την πρόταση. Βέβαια, είναι κάπως ανησυχητικό ότι πολύ τολμηρές προτάσεις αμφισβητούνται είτε στο Συμβούλιο είτε στο Κοινοβούλιο. Οπότε θα ήθελα να καλέσω και τη δική σας Επιτροπή να έχει και μια πιο οριζόντια προσέγγιση και να δει τι συμβαίνει στις ε, συγκεκριμένες επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στην Επιτροπή, Περιφερειό, στην ε, Επιτροπή Περιφερειακών Θεμάτων, ε, την Επιτροπή Γεωργίας, γιατί σε αυτές τις επιτροπές γίνονται οι διαπραγματεύσεις για ζητήματα τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά για τις μελλοντικές διαδικασίες χορήγησης απαλλαγής. Θα ήθελα επίσης ε, να αναφερθώ και στα ερωτήματα ε, ε, του κυρίου Μούλτερ και τα σχόλιά του σε σχέση με τις τις προαιρετικές δηλώσεις και τις ετήσιες συνόψεις. Αποφασίσαμε με, τις, με τους συνομοθέτες, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο, για το θέμα ε, του δημοσιονομικού κανονισμού που συμπεριλαμβάνει αυτά τα τρία στοιχεία και τον ενισχυμένο ρόλο των ε, ετήσιων συνόψεων, όπως επίσης και μία δήλωση διαχείρισης. Ε, τα έγγραφα αυτά μάλιστα θα είναι αντικείμενο ανεξάρτητου ελέγχου και θα ήθελα τώρα να αναφερθώ και στο ερώτημα του κυρίου Οντί στις ε, συναντήσεις ε, που έχω στα κράτη-μέλη, προσπαθώ πάντοτε να βλέπω, να συναντώ τα ανώτατα όργανα ελέγχου και να τα πείσω ότι εκείνα πρέπει να αναλάβουν ε, τις ετήσιες συνόψεις και τις δηλώσεις διαχείρισης γιατί γνωρίζουν καλύτερα την κατάσταση στο δημόσιο τομέα και συνεπώς αυτό θα βοηθά την συνοχή του συνολικού ελέγχου, αλλά φυσικά δεν μπορούμε να τους επιβάλλουμε να το κάνουν λόγω της ανεξαρτησίας τους. Επομένως, έτσι έχουν τα πράγματα αυτή τη στιγμή. Όσον αφορά τώρα το ειδικό ερώτημα του κυρίου Μόλτερ σε σχέση με τα καρότα που μπορούμε να προτείνουμε, για την ευρύτερη εισαγωγή, για την ευρύτερη αποδοχή ε, των γραπτών δηλώσεων, να σας πω. Πρώτον, πρέπει να δούμε το σύστημα της ε, δήλωσης διαχείρισης πώς λειτουργεί, γιατί πρέπει να αναπτύξουμε όλους τους απαραίτητους κανόνες για το πώς πρέπει να συμπληρώνονται αυτές οι γραπτές ε, δηλώσεις. και παράλληλα να αρχίσουμε συζητήσεις με τα κράτη-μέλη για την ευρύτερη εφαρμογή πολιτικών δηλώσεων. Τώρα προβληματιζόμαστε σε σχέση με το πώς να καταστήσουμε πιο ελκυστικές αυτές τις ε, δηλώσεις γραπτές. Βέβαια είναι πρόημο να πει κανείς ότι υπάρχει μια συγκεκριμένη συνταγή γι' αυτό, αλλά σε κάποιους τομείς ε, έχουμε Αντίστοιχε εξελίξεις. Για παράδειγμα, στον τομέα των τελωνίων έχουμε το σύστημα του εγκεκριμένου οικονομικού ε, φορέα, που σημαίνει ότι αν μία ε, εταιρεία πληρεί κάποιες προποθέσει υπόκειται σε λιγότερους ελέγχους ε, τελωνιακή φύσεως. Τα καρότα λοιπόν στα οποία αναφέρομαι ε, αφορούν τη συγκεκριμένη ε, προσέγγιση. Μπορεί όμως αυτό να αποτελέσει και αντικείμενο συζήτησης μεταξύ Κοινοβουλίου και Επιτροπής και φυσικά είναι κοινός μας στόχος να έχουμε αυτές τις ε, θελοντικές δηλώσεις οι οποίες θα πρέπει να γίνουν αποδεκτές στα κράτη-μέλη. Μετά υπάρχει το θέμα της συγκρισιμότητας ε, των ε, ποσοστών σφαλμάτων, το οποίο το έθεσε ο κύριος Πίπερ. Ενδεχομένως, να πρέπει να απευθύνει το ερώτημά σα στο ελεκτικό συνέδριο, γιατί είναι δικός του ρόλος ε, η εξασφάλιση της συγκρισιμότητας των στοιχείων. Ελπίζω να, μπορούν, να μπορέσουν να το εξηγήσουν να εξηγήσουν τι προτίθενται να κάνουν σε αυτή την περίπτωση. Γιατί είναι γεγονός ότι ειδικότερα από το επόμενο έτος, όπως πολύ σωστά το είπε και ο κύριος Γκάιερ, η μεθοδολογία του ελεγκτικού συνεδρίου θα αλλάξει και επομένω είναι πάρα πολύ σημαντικό να εξασφαλίσουμε ότι τα νέα στοιχεία τα οποία θα παρέχονται, θα, θα, θα, παρασχεθούν για την απαλλαγή του 2013 να είναι συγκρίσιμα με αυτά των προηγούμενων ετών. Αλλά αυτό βέβαια πρέπει να μας το εξασφαλίσει το ελεγκτικό συνέδριο. Όσον αφορά τώρα το θέμα των αξιοπίνων πράξεων ε, στα κράτη-μέλη, δηλαδή ότι η Εγκληματίε ε, χρησιμοποιούν τις πιο δύναμες δομέ στα κράτη-μέλη. Ναι, αυτό έχει να κάνει με την μελέτη αξιολόγησης αντικτύπου, η οποία συντάχθηκε όταν προετοιμάσαμε την ε, πρότασή μα για την Οδηγία Προστασίας των Οικονομικών Συμφερόντων. Η οδηγία αυτή είναι ουσιαστικά απάντηση σε αυτή την κατάσταση, μια αντίδραση, γιατί προσπαθήσαμε, να προσπαθήσαμε έτσι να εναρμονίσουμε την αντιμετώπιση των ε, εγκληματικών πράξεων ε, ή τέλος πάντων των απατών που ε, θα μπορούσαν να είναι αντικείμενο κυρώσεων. Υπάρχουν βέβαια ελάχιστες και μέγιστες κυρώσεις και υπήρχαν και πολλά άλλα μέτρα που θα επιτρέψουν την εναρμόνιση της ποινική νομοθεσίας σε σχέση με την προστασία των ε, ενωσιακών ε, οικονομικών συμφερόντων. Και θα ήθελα να σας ε, καλέσω προκειμένου να ορίσετε να εισηγητή για αυτό το πολύ σημαντικό θέμα, αυτή την πολύ σημαντική πρόταση, γιατί έχει αρχίσει ήδη η συζήτηση στο Συμβούλιο και και υπάρχουν πολύ αντιφατικέ απόψει. καταρχάς σε σχέση με την νομική βάση για την πρόταση αυτή. Η νομική βάση είναι πάρα πολύ σημαντική. Γιατί οι συνομοθέτες ε, αν αποφασίσουν να δεχθούν τη νομική βάση που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τότε όλα τα κράτη-μέλη θα είναι σε ισότιμη βάση. Αν επιλεγεί μια άλλη, κράτη, μια άλλη νομική βάση, τα τρία κράτη-μέλη που ήδη υποστηρίζουν την άποψη αυτή, το Ηνωμένο Βασίλειο δηλαδή, η Ιρλανδία και η Γερμανία, θα είχαν opt-out από την νομοθεσία αυτή. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι η νομοθεσία αυτή, αν τα κρατημέλη όντω ε, επιλέξουν να μην συμμετέχουν, επιλέξουν το opt-out, θα ισχύει για 24 και όχι για 27 κρατημέλη. Άρα, περνάω στο επόμενο ερώτημα του κυρίου Σκυλακάκη. Έθεσε το θέμα της, ε, των ερευνών ιδίας πρωτοβουλίας. Εγώ δεν βλέπω την αντίφαση ανάμεσα στη δική μου απάντηση τον Νοέμβριο και της ε, γραπτής μας απάντησης. Ε, αυτό που προσπαθήσαμε να πούμε είναι ότι δεν θεωρούμε ότι οι έρευνες που λαμβάνουν χώρα βάση πληροφοριών τρίτων μερών πρέπει να αντιμετωπίζονται ως ε, παθητική δράση. Αντιθέτως, όλα αυτά που συζητήσαμε σε σχέση με το whistleblowing στην, ε, και στην Επιτροπή σας αποκάλυψαν πόσο σημαντικό είναι να εξασφαλίσουμε τη, τους σωστούς όρους για αυτούς οι οποίοι μας ενημερώνουν για ενδεχόμενες παρατυπίες να μπορούν να γνωστοποιήσουν τα πορίσματά τους στις αρχές, ώστε να μπορούν αυτές να αναλάβουν δράση. Άρα εξακολουθώ να συμφωνώ μαζί σας ότι πρέπει να ενισχύσουμε την ε, δυνατότητα ερευνών ιδίας πρωτοβουλίας. Πολύς προσφάτως μάλιστα ορίσαμε ένα νέο γενικό διευθυντή ένα νέο διευθυντή, ο οποίος είναι υπεύθυνο για τις εσωτερικές ε, έρευνες. Και έχουμε γενικώ αρκετούς νέους διευθυντές, οπότε πιστεύω ότι αυτές οι νέες δυνάμεις θα επιτρέψουν εύλογη προσοχή στις ε, έρευνες αυτές ίδιας πρωτοβουλίας εγώ θα ήθελα να υπάρχει στενότερη σχέση μεταξύ των εσωτερικών ελέγχων και της Όλαφ ως προς τη χρήση των πληροφοριών ε, των ε, εσωτερικών ε, ελεγκτικών αρχών με πολύ πιο αποτελεσματικό τρόπο στις έρευνες. Όσον αφορά τώρα τι ερωτήσει του κυρίου Στάις και τις ειδικέ εκθέσεις, έχουμε μια πάρα πολύ σαφή διαδικασία για τις ειδικέ εκθέσεις και Υπάρχει μια κεντρική υπηρεσία η γενική, στη Γενική Διεύθυνση προπολογισμών, ε, που έχει μια βάση δεδομένων όλων των συστάσεων ε, που ε, υποβάλλονται από το ελεγκτικό συνέδριο. Υπάρχει λοιπόν πολύ διεξοδική παρακολούθηση αυτών των συστάσεων και βέβαια η υπηρεσία που είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή είναι η υπηρεσία από την οποία η οποία έχει καταγράψει αυτές τις συστάσεις. Με την παρακολούθηση αυτή, αν κάτι δεν πάει καλά ή αν υπάρχουν καθυστερήσεις, τότε συζητούμε αυτό το θέμα στην Επιτροπή ε, Ελέγχου ε, ή εγώ στέλνω ας πούμε επιστολές ε, στους ε, υπόλοιπους συναδέλφους της Επιτροπής για την, σε σχέση με την καθυστέρηση της μίας ή της άλλης σύστασης. Έχουμε δηλαδή πάρα πολύ συγκεκριμένη αυστηρή διαδικασία ως προς αυτό. Όσον αφορά τώρα το ερώτημα της χορήγησης απαλλαγής στο Συμβούλιο και τη δική μου θέση. Νομίζω ότι εγγράφως ε, την ε, παρουσίασα τη θέση μου και τη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εξακολουθούμε να θεωρούμε ότι οι υπάρχουσες ε, διατάξεις της συνθήκης και η εφαρμοστική νομοθεσία μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε απαλλαγή και στο Συμβούλιο ε, και, στην Επιτροπή. Βέβαια, πρέπει να καταλάβετε ότι είμαι σε λίγο δύσκολη θέση για να δώσω πολύ συγκεκριμένες συμβουλές για αυτό το θέμα. Αλλά το συζητήσαμε με την κυρία Γιάλα Σέντερ ε, πολλές φορές. Ποιος θα μπορούσε δηλαδή να είναι ο τρόπος ε, να επιφέρουμε σοβαρές αλλαγές σε αυτό το θέμα. Δεν είναι πολύ απλό νομίζω εγώ. να μεταφέρεται απλώς ε, η απαλλαγή ε, στην Επιτροπή, γιατί αν εμείς είμαστε υπεύθυνοι, τότε θα πρέπει να λάβουμε όλες τις πληροφορίες και να έχουμε και πλήρη πρόσβαση στα ε, έγγραφα του Συμβουλίου, κάτι το οποίο βέβαια δεν είναι προς συμφέρον του Συμβουλίου, το να παρέμβουμε δηλαδή τόσο πολύ σε αυτά που κάνει το Συμβούλιο. Νομίζω λοιπόν ότι η διαδικασία που έχει ακολουθηθεί τα τελευταία δέκα χρόνια, ίσως και παραπάνω, θα πρέπει να συνεχίσει και πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να βγούμε από αυτό το διέξοδο. Όσον αφορά τώρα την ενημέρωση από την Όλαφ που ζητήσατε για τις συμφωνίες για τα καπνά. Η κατάσταση έχει ως εξής. Μόλις διευκρινίσατε, μόλις τι θέλατε από, να σας ε, γνωστοποιήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επιλέξαμε κάποια στοιχεία και σας τα υποβάλαμε στο Κοινοβούλιο. Τώρα, αν υπάρχει ακόμη έλλειψη πληροφοριών, εμείς ε, ευχαρίστως ε, να ε, σας δώσουμε και τις υπόλοιπες απαραίτητες πληροφορίες. Δεν έχουμε και τίποτα να κρύψουμε εμείς αυτή την υπόθεση. Είμαστε πλήρως διαφανείς. Όσον αφορά το θέμα του Επιτρόπου Ντάλι, θα ήθελα να είμαι σαφής. Ο κύριος Στάις σε αυτό το θέμα είπε ότι είμαι υπεύθυνο και για την Όλαφ. Ε, είναι όμως σημαντικό να συμφωνήσουμε όλοι ότι το ερευνητικό τμήμα της Όλαφ πρέπει να γίνεται, πρέπει να διεξάγεται ανεξάρτητα. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό για να εξασφαλίσουμε ότι η Όλαφ δεν θα αρχίσει ε, να, να, να ε, ε, αναμειγνύεται σε πολιτικές συγκρούσεις κλπ. κλπ. Αυτό ήταν βασικό τμήμα της νομοθεσίας, στην οποία τελικά καταλήξαμε με το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Χάρη στις προσπάθειες κυρίας Γκρέσλε και της καλές προσπάθειες των ε, Προεδριών του Συμβουλίου. Ελπίζουμε να εγκριθεί σύντομα η σχετική νομοθεσία. Από ό,τι κατάλαβα, η Προεδρία έχει βρει μια λύση σε σχέση με την πρόσφαση στις πληροφορίες. Οι νομικές υπηρεσίες τώρα των ε, δύο οργάνων ε, ασχολούνται με την επεξεργασία των πληροφοριών που χρειάζονται και ελπίζω να επιληθεί το ζήτημα. Είναι πολύ σημαντικό να μην Είναι πολύ σημαντικό να έχουν τη δυνατότητα οι εθνικές εποπτικές αρχές να ασχολούνται με τα θέματα αυτά, γιατί ουσιαστικά ε, για εθνικό ζήτημα πρόκειται. Όσον αφορά τώρα το θέμα του κυρίου Πετή, ως μέλους της Επιτροπής, δεν ήταν ουσιαστικά ορισμός, ήταν ε, εκ νέου ορισμός ολόκληρης της Επιτροπής και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είχε κανέναν ιδιαίτερο λόγο να αμφισβητήσει τον ορισμό αυτό, γιατί αυτό δεν είναι λομπίστας, είναι νομικό σύμβουλος σε αυτή τη συγκεκριμένη εταιρεία. Και αν δούμε το ιστορικό των δραστηριοτήτων του, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν βλέπει να υπάρχει κανένα πρόβλημα και επειδή λαμβάνεται υπόψη βέβαια και ε, η ε, προηγούμενη του εμπειρία ως ε, επικεφαλής νομικής υπηρεσίας, νομίζω ότι στην Επιτροπή Δεοντολογίας είναι ένας πολύ σημαντικός άνθρωπος, γιατί ακριβώς γνωρίζει τι γίνεται. Και αυτό σας το λέω απαντώντας στο ερώτημά σας για το πώς βλέπουμε εμείς αυτό το θέμα στην Επιτροπή. όσον αφορά τον Όλαφ και την ε, ποπτική Επιτροπή. Δεν πρέπει να μας διαφεύγει ότι η Εποπτική Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την εποπτεία και των ανακρίσεων της Όλαφ Γι' αυτό ακριβώς την έχουμε ε, αυτή την Επιτροπή, είναι για να μην υπάρχει πολιτική παρέμβαση. Γι' αυτό πιστεύω ότι η Εποπτική Επιτροπή πρέπει να, συνεργάζεται, πρέπει να συνεργάζεται με την Όλαφ για να μπορέσει να βρει λύσεις αν υπάρχουν προβλήματα. αλλά θα ήθελα να επαναλάβω το εξή ότι συνεργάζομαι πολύ με την Όλαφ σε θέματα πολιτικών και για την προετοιμασία της στρατηγικής καταπολέμησης της απάτης, αλλά και για την εφαρμογή της στρατηγικής καταπολέμησης της απάτης. Ο κανονισμός της Όλαφ και οι υπόλοιποι κανόνες ε, με παρεμποδίζουν από παρέμβαση ε, στις ανακριτικές ε, δραστηριότητες της Όλαφ και νομίζω, θέλω να επαναλάβω δηλαδή ότι αυτό είναι προς όφελος όλων. Νομίζω ότι απάντησα σε όλα τα ερωτήματα που μου απευθύνατε. Αυτά λοιπόν. Κύριε Πίτροπε, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Ε, ότι όσο ο Επίτροπος Αρμόδιος για την Όλαφ ε, δεν μπορείτε να εμπλακείτε κι εσείς στις ανακρίσεις, ε, πρέπει να υπάρχει κάποια αμεροληψία και κάποια ανεξαρτησία. Όταν όμως η Επιτροπή Ελέγχου λέει ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα στις ανακρίσεις και εφόσον η έκθεση αυτή φτάσει στον ε, διευθυντή της Όλαφ, και από την έκθεση αυτή εξαχθούν κάποια συμπεράσματα, τότε θα πρέπει και εσείς ως Επίτροπος να μπορείτε να αντιδράσετε. Δηλαδή η Επιτροπή Ελέγχου λέει ότι υπάρχουν ίσως ε, κάποια προβλήματα. Ε, ασχολείται με αυτά ο διευθυντής της Όλαφ, άρα και εσείς έχετε να παίξετε κάποιο ρόλο. Κοιτάξτε, το θέμα του ότι είμαι επίτροπος ε, αρμόδιος για την Όλαφ αυτό σημαίνει ότι είμαι αρμόδιος για την πολιτική καθοδήγηση και για τις πολιτικές δραστηριότητες της ε, Όλαφ. Αυτά που μόλις τώρα εσείς είπατε, ε, απλά ε, παίρνουν το μέρος ή της, της μίας ή της άλλης πλευράς δεν πρέπει να υπάρχει πολιτική παρέμβαση και μπορείτε να δείτε ας πούμε στο δικαστήριο στο Στρασβούργο πόσες ε, περιπτώσεις που παραπέμπονται στο δικαστήριο του Στρασβούργου τελικά επιλύονται με πολιτική παρέμβαση στην όλη διαδικασία. Εγώ λοιπόν έχω σαφή άποψη επί του θέματος. Τώρα τρέχει η ε, δικαστική διαδικασία και είμαι σίγουρος ότι η πολιτική παρέμβαση απλά θα ζημιώσει την διαδικασία που έχει ξεκινήσει έτσι και αλλιώς. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Επίτροπε. Άλλοι δύο συνάδελφοι και έχουμε και άλλα δύο θέματα. Όλα αυτά πρέπει να τα κάνουμε σε 30 λεπτά. Ε, και αν μπορείτε να μου υποσχεθείτε ότι ε, θα τα καταφέρουμε, Πολύ ωραία. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Μούλντορ, στην κυρία Πίπερ, μετά στον ε, ε, ε, ελεγκτικό συνέδριο. Κοιτάξτε, εγώ απογοητεύτηκα. Είναι απογοητευτικό το γεγονός ότι μετά από τόσα χρόνια η Κομισιόν εξακολουθεί να μην ε, γνωρίζει πώς πρέπει να ε, υλοποιεί τις απόψεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σε αυτή τη φάση, έχοντας δει τώρα ψηφίσματα για 10 περίπου χρόνια, νομίζω ότι η κατάσταση είναι ιδιαίτερα απογοητευτική. Εμείς λοιπόν, στο πλαίσιο της διαδικασίας απαλλαγής, ε, θα προσπαθήσουμε να δούμε πώς μπορεί να αλλάξει η άποψη της Επιτροπής. Ευχαριστούμε πολύ που κρατήσατε το χρόνο του ενός λεπτού και η κυρία Πίπερ, ο κύριος Πίπερ με συγχωρείτε. Ε, κύριε Επίτροπε, και εγώ δεν είμαι ιδιαίτερα ευχαριστημένος. Ε, καταρχήν όσον αφορά τη συγκρισιμότητα των δεδομένων και των ποσοστών σφάλματος. Ε, αυτά που είπαμε δεν αφορούν μόνο το ελεγκτικό συνέδριο, αλλά κυρίως την Κομισιόν. Δηλαδή, ε, σχετικά με τη συγκρισιμότητα εκτέσεων, ελέγχων γεωργικής, διαρθρωτικής πολιτικής, ερευνητικής πολιτικής. Ε, δεν πρέπει ο ένας να πετάει τον μπαλάκι στον άλλον, αλλά μέσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εντοπιστεί ποιοι τομεί λειτουργούν με τον βέλτιστο τρόπο. Κατόπιν, για την έκθεση όλα. Κοιτάξτε, σε όλες τις δημοκρατίες έχουμε κοινοβούλια τα οποία με έμπιστους ανθρώπους στον τομέα της άμυνας, της καταπολέμησης απάτης, ε, έχουν δικαίωμα να εκφράζουν τα άποψή τους. Το θέμα δεν είναι να χαράσουν πολιτική. Γι' αυτό λοιπόν σας ερωτώ ξεκάθαρα. Εσείς γιατί έχετε τόσο μεγάλο πρόβλημα να επιλέξετε έναν έμπιστό σας από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να το συμπεριλάβετε στην ενημέρωση. Μήπως έχετε τίποτα να κρύψετε. Πρόεδρος, πολύ ωραία. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στην κυρία Καγιολάιτ, στην εκπρόσωπο του ελεγκτικού συνεδρίου που ζητάει το λόγο εδώ και πολύ ώρα για το θέμα της μεθόδου. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ο κύριος Πάιπερ, κύριε Ανδρέας και άλλοι ε, έκαναν ε, μία σαφή ερώτηση. Ε, τι γίνεται τελικά με τις συναλλαγές και νομίζω ο κύριος Κόγερ είχε την απάντηση στην ομιλία του. Μίλησε για την αντικατάσταση. Το κόστος του να δικαιολογήσει κανείς ένα είναι πολύ χαμηλό ενώ τα χρήματα όμως ε, χάνονται και αν δεν αλλάξουμε δεν θα αλλάξει τίποτα. Έρχομαι τώρα στην μεθοδολογία του δικαστηρίου. Ο κύριος Επίπε και ο κύριος Γκάιερ έκαναν μια έκκληση να σταθεροποιήσει το ε, δικαστήριο, το ελεγκτικό συνέδριο τη μέθοδο όταν υπολογίζει το σφάλμα υπολογίζεται το σφάλμα και για τη συγκρισιμότητα το κάναμε για την cross compliance ε, δυστυχώς όμως ο κύριος Κάιερ είπε ότι είναι δικαίωμα του δικαστηρίου, του ελεγκτικού συνεδρίου να αλλάξει τη μέθοδο. Εγώ θα έλεγα είναι περισσότερο υποχρέωσή του. Και όσον αφορά τη σταθερότητα, η σταθερότητα δεν μπορεί να εγγυήσει, ε, να, να εγγυηθεί την ε, πραγματική βελτίωση. Συγκεκριμένα, το 2011 τα λάθη της πολλαπλούς ε, συμμόρφωσης ε, μετρήθηκαν ποσοτικά γιατί διαπιστώθηκε ότι το ε, ελεγκτικό συνέδριο δεν επηρέασε καθόλου το λάθος ήταν στο 0,1 στο σύνολο του πληθυσμού. Επίσης, όσον αφορά τις προκαταβολές, αυτές αφαιρούνται από το ελεγκτικό συνέδριο και δεν συνδυάζονται τόσο με την συνοχή και τις ε, προκαταβολές. Αυτά ποτέ δεν ε, συμπεριλαμβάνονταν στους ελέγχους του ε, ελεγκτικού συνεδρίου. Άρα δηλαδή η αλλαγή δεν είναι μεγάλη και η αλλαγή αυτή επουδενή δεν θα αυξήσει τα ποσοστά σφάλματος και δεν αλλάζει το ε, ελεγκτικό συνέδριο τους κανόνες, απλά αλλάζει τις διακυμάνσεις, γιατί μπορεί να αλλάξει και όγκος των προκαταβολών. Στην αρχή της περίοδου είναι υψηλές οι προκαταβολές και μετά σιγά σιγά μειώνονται. Αυτό μπορεί να δίνει την εντύπωση ότι αυξάνονται, μειώνονται τα ποσοστά λάθους, αλλά αυτά δεν ισχύουν. Επίσης, ε, όσον αφορά τη συγκρισιμότητα, αυτή υπάρχει ε, τα τελευταία χρόνια, ισχύει ε, στα ε, τυπικά λάθη, όπως ακριβώς διαπιστώθηκε στο επίπεδο σημαντικότητας. Επίσης, για το 2011 η Κομισιόν όταν έδωσε τις οδηγίες για το πώς θα υπολογίζεται το υπολοιπόμενο ποσοστό λάθους, Εκεί θέλω να σας πω, εδώ θέλω να σας πω ότι εμείς δεν κάνουμε, δεν δημιουργούμε νέους κανόνες, απλά ακολουθούμε αυτά που έχουν αποφασιστεί. Το τελευταίο που αναφέρθηκε ήταν η συγκρισιμότητα του σφάλματος μεταξύ στην ε, Κομισιόν και το Ελεγκτικό Συνέδριο σχετικά με τις, ε, τις ε, δημοκρατικές, τις δημόσιες αναθέσεις έχει υπολογιστεί το ποστό σφάλματος για το σύνολο του προϋπολογισμού και η μέθοδος ε, συγκρίθηκε με διάφορες γενικές διευθύνσεις, ε, παρέμοντας χάρη αυτή την, ε, των περιφερειών. Επίσης, αναφέρθηκε τουλάχιστον στην αγγλική μετάφραση ότι κάθε λάθος είναι λάθος 100% αυτό όμως δεν είναι αλήθεια Ε, αλλάζει ο σκοπός ε, ακόμα και αν τα σφάλματα οδηγούν στο να κατακαιρωθεί ο διαγωνισμός σε λάθος δικαιούχο. Ακόμα και εκεί και σε αυτές τις περιπτώσεις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, δεν το υπολογίζει ως 100% λάθος. Σε άλλες περιπτώσεις όπου το συνέδριο λέει λάθος 100% η Κομισιόν μπορεί να είναι πιο κάτω και όταν το ε, συνέδριο έχει μηδέν σφάλμα, τότε μπορεί η Κομισιόν να έχει ε, ποσοτικό ε, σφάλμα. Γι' αυτό λοιπόν έγιναν συγκρίσεις και οι διαφορές είναι πολύ μικρές και οι διαφορές εξηγούνται, μπορούν να εξηγηθούν και οι δύο πλευρές τις έχουν αποδεχτεί γιατί σε τελική ανάλυση δεν οδηγούν σε μεγάλη διαφορά στο τελικό αποτέλεσμα. Ο κύριος ρώτησε κατά πόσον η δήλωση αξιοπιστίας μπορεί να είναι σαφέστερη διότι το δικαστήριο ε, τοποθετηθείται θετικά στους λογαριασμούς και αρνητικά στις ε, πληρωμές. Αυτό είναι αλήθεια. Ε, τα διεθνή λογιστικά πρότυπα λαμβάνουν υπόψη τους μια κατάσταση όπου πρέπει κανείς να συμβιβάσει αποτελέσματα δύο διαφορετικών ελέγχων. με βάση την ε, ισχύουσα νομοθεσία προκύπτουν λάθη στις δαπάνες. Κατόπιν τούτου, ε, κάτω από το, από το πρίσμα της ε, τακτικότητας, είναι αρνητικό το αποτέλεσμα. Το θέμα όμως είναι ότι αυτά απορρέουν από τη συνθήκη όπου αναφέρεται ότι το συνέδριο πρέπει να τοποθετηθείτε σχετικά με, την, με τον τρόπο που γίνονται οι λογαριασμοί. Θα ήθελα να επισημάνω και κάτι άλλο στο σχόλιο του κυρίου Μούλντερ σχετικά με τις δηλώσεις αξιοπιστίας. Το συνέδριο θέλει να πει ότι ανεξάρτητα με το κατά πόσο μία δήλωση είναι υποχρεωτική ή δεσμευτική, ακόμα και τώρα υπάρχουν πολλές δηλώσεις που περιλαμβάνουν ποσοστά σφάλματος. Εμείς πιστεύουμε είναι πολύ σημαντικό σε όλες αυτές τις περιπτώσεις τα δεδομένα πάνω στα οποία βασίζονται οι δηλώσεις αξιοπιστίας να είναι διαφανή, να είναι κατανοητά στην Κομισιόν, στο Κοινοβούλιο και ίσως και στην ελεγκτική αρχή. Πώς δηλαδή γίνεται η δήλωση προς την Κομισιόν. Μόνο έτσι έχει νόημα η δήλωση αξιοπιστίας και μόνο έτσι μπορούμε να περιμένουμε ότι κάποια στιγμή θα μπορεί κανείς και να βασιστεί σε αυτές τις δηλώσεις. Σας ευχαριστούμε πολύ κυρία Καλιουλάιτ για αυτές τις ε, διευκρινήσεις. Και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στον Επίτροπο Σεμέτα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ δυνατόν για μια σύντομη απάντηση. Θα είμαι σύντομος, ε, θα απαντήσω στον κύριο Μίλντερ. Νομίζω πως πρέπει να κατανοήσουμε ότι κάναμε ένα μεγάλο επίτευγμα με την έγκριση των διατάξεων για τις δηλώσεις ε, διαχείρισης αλλά και τις εθνικές δηλώσεις στο πλαίσιο του δημοσιονομικού κανονισμού. Ε, θα θυμίσετε σίγουρα το πόσο δύσκολο ήταν αυτό το έργο και όπως είπε η κυρία Καλωραϊτ αυτό που είναι το πιο σημαντικό είναι οι πληροφορίες οι οποίες τροφοδοτούν αυτές τις δηλώσεις θα πρέπει να είναι αξιοπιστές. Και θα πρέπει πρώτα να διασφαλίσουμε ότι αυτές οι πληροφορίες ε, στις ε, δηλώσεις διαχείρισης είναι αξιόπιστες. Γι' αυτό και οι υπηρεσίε μας δουλεύουν πάνω σε αυτό. Αυτή, αυτό το θέμα της εθελούσιας δήλωσης ε, είναι το προσεχές βήμα, το επόμενο βήμα και έχω πει επαντηλημένη κατά διάρκεια της διαδικασίας απαλλαγής Πιστεύω πως και πολιτική ευθύνη για θέματα λογοδοσίας είναι κάτι το οποίο θα μας βοηθήσει, αλλά θα πρέπει να θέσουμε τις σωστές βάσεις και είμαστε τεθειμένοι να συνεργαστούμε με το Κοινοβούλιο σχετικά με την εξέβρεση λύσης. Τώρα για πρόσβαση στις πληροφορίες, στην υπόθεση Νταλή, <clears throat> να επανελάβω πως βρέθηκε τρόπος ε, συνεργασίας μεταξύ των δύο οργάνων και οι νομικές υπηρεσίες των δύο θεσμικών οργάνων εξετάζουν τα έγγραφα και θα καταστήσουν διαθέσιμα έτσι ώστε όσοι το Κοινοβούλιο επιθυμούν μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτές τις προφορίες. Και ο πρόεδρος είναι αυτά τα πρόσωπα που επιθυμούν να λάβουν τις προφορίες αυτές. Τώρα, σε ό,τι φορά τη συγκρισιμότητα των προφοριών που προέρχονται από διάφορες γενικές διευθύνσεις, τα προηγούμενα δύο έτη ασχοληθήκαμε ιδιαίτερα με την περαιτέρω εξέλιξη των μεθοδολογιών σε εκθέσεις ε, λειτουργικότητας ε, και θέλαμε να διασφαλίσουμε καλύτερη συνοχή, συνέπεια και συγκρισιμότητα ανάμεσα στις εκθέσεις, ε, τις εκθέσεις των γενικών διευθύνσεων το 2011 για πρώτη φορά συμπεριλάβαμε τον ορισμό του εναπμένοντος ποσοστού σφάλματος και σε αυτή τη διαδικασία απαλλαγής έχουμε διαφορετικές διαδικασίες προόδου για τον καθορισμό του επίπεδου σφάλματος και εξετάζουμε την καλύτερη και πιο στενή δυνατότητα συγκρισιμότητας ε, μεταξύ των τετήσεων εξέσεων της ε, Επιτροπής. Αν δείτε την ε, έκθεση δραστηριοτήτων του 2011 και τα βρήματα του ελεγχτικού συνεδρίου δεν υπάρχουν πολλές διαφορές όπως το συνέβαινε στο παρελθόν. Λοιπόν, όλο και πλησιάζουμε, όλο και προσεγγίζουμε να αποκτήσουμε μια κοινή γλώσσα ανάμεσα στην Κομισιόν και το Ελεκτικό Συνέδριο. Και αυτό έχει μεγάλη σημασία. Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε το... Θα σας ευχαριστήσω, Επίτροπε, σε μέτα για το ότι πετύχατε τον προηγούμενους μήνες ε, εντάξει, ασχήθηκαν κάποιες ε, κριτικές, ε, δικαιολογημένες, θεμητέ, αλλά θα θέλαμε να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Σας ευχαριστώ που βρεθήκατε ανάμεσά μα και απαντήσατε στι ερωτήσει. Θα δώσω το λόγο στον εισηγητή, αν επιθυμεί να τον λάβει. Κοιτάξτε, θα έλεγα να προχωρήσουμε στην ημερήσια διάταξη. Είχαμε μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση και υπάρχουν εδώ συνάδελφοι ε, που επιθυμούν να συζητήσουν για το επόμενο θέμα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Επίτροπε, και τα ξαναλέμε. liebe Kollegen und Kollegen, äh, ich die Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, εγώ καθυστέρησα να έρθω. Ε, έχουμε όμως τώρα ένα θέμα το οποίο πρέπει οπωσδήποτε να το συζητήσουμε. Βέβαια οι διερμηνείς ε, θα παραμείνουν κοντά μας μέχρι τις 6.30 και εάν δείξουμε πειθαρχία θα τα καταφέρουμε με το επόμενο θέμα. Πρόκειται για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης ε, και θα ήθελα να καλωσορίσω τον κύριο Τάμσιν Μπάουτεν Γενικό Διευθυντή για Ενέργειες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προέρχεται από την Τράπεζα Επενδύσεων του Λουξεμβούργου. Και χαίρομαι πάρα πολύ που είσαστε εδώ. Ο ε, εισηγητής είναι ο κύριος Σόρεν Σόντεργαρτ, τον οποίο και ε, παρακαλώ να μας εισαγάγει στο θέμα όσο πιο σύντομα γίνεται. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τις απαντήσεις στα 24 ερωτήματα που θέσαμε και συγχρόνως να ευχαριστήσω και την εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων που βρίσκεται ανάμεσά μας σήμερα. Δεν νομίζω ότι αλλάζουν πολλά πράγματα από την αρχική μας θέση. Είναι κάτι το οποίο εξτάσαμε παντελημένως. Η Τράπεζα Επενδύσεων και οι διευκολύνσεις της ε, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στο πλαίσιο της διαδικασίας απαλλαγής. Ξέρετε τι συνέβη στο ε, πλαίσιο του Κοτονού και ελπίζω η εκπρόσωπος τη Ευρωπαϊκή Τράπεζας Επενδύσεων θα εγκρίνουν την τροποποίηση που προτείνουμε. Και έχω 7 ερωτήσεις. 7 ερωτήσει συγκεκριμένε, σαφείς, μετά από τι απαντήσει που ήδη λάβαμε. Καταρχήν, η ΕΤΕ βρίσκεται στην 37η θέση επί 58 σε ό,τι αφορά τον δείκτη διαφάνειας. μακριά από την Ευρωπαϊκή, με την Διεθνή Τράπεζα. Η ΕΤΕ συχνά έχει πολλές ε, υποχρεώσεις. Ε, Δεδομένου όμως ότι πρόκειται για δημόσια κονδύλια τα οποία διαχειρίζεται, θα ήθελα η τράπεζα να μας δώσει κάποια παραδείγματα για να γνωρίζουμε τι ακριβώς συμβαίνει αναφορικά με αυτές τις εμπιστευτικές ε, δεσμεύσεις. Επίσης, θέλαμε κάποια στοιχεία που θα βελτίωναν την διαφάνεια σε ό,τι φορά τις τραπεζικές τις δραστηριότητες και στις ερωτήσεις μας φυσικά προσπαθήσαμε να βρούμε τι ακριβώς συμβαίνει με τους φορολογικούς παραδείσους και τα ποσά τα οποία αναφέρονται εδώ είναι τεράστια. Η τράπεζα δήλωσε ότι καταβάλει κάθε προσπάθεια για να αποφύγει αυτές τις τάσεις. ότι έλειψαν κάποια μέτρα, η τράπεζα δεν μπορεί να αποκλείσει ότι μπορούν ε, να γίνουν κάποιες μεταφορές ε, κονδυλίων στους φορολογικούς προς τους φορολογικούς παραδείσους. Θα ήθελα λοιπόν να ζητήσω από την τράπεζα κατά πόσο θα μπορούσε να μας πει ποιες είναι οι χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης που δημιουργούν προβλήματα σε θέματα τραπεζικών απορρίτων. Και κάτι ακόμα, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι οι περιπτώσεις στις οποίες εμπλέκεται και η Κομισιόν και κατά πόσον υπήρξε μια σημαντική αύξηση την περίοδο 2009-2011. Και με βάση όλα αυτά θέλω να μάθω σε τι οφείλεται αυτή η αύξηση. Θα να γνωρίζω εάν είχαμε τέτοια αποτελέσματα, εάν είχαμε πάρει μια ψαλίδα χρονική ευρύτερη. Εδώ μιλάμε για mainstreaming σε θέματα ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θα θέλω να μάθω ποιε είναι οι τροποποιήσεις, ε, οι αλλαγές ε, στις οποίες θα μπορούσε να αναφερθεί και θα μπορούσαμε να έχουμε τι δραστηριότητε και τα αποτελέσματα αυτών σε ζητήματα mainstreaming. Ζητήσαμε από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να δημοσιεύσει έναν πίνακα με τους ε, μισθούς ε, μας είπαν ότι εκπροσωπούν, αντιπροσωπούν το 16% και εγώ πιστεύω ότι τα στοιχεία που μας ε, δώσατε δεν είναι επαρκή. Θέλαμε να γνωρίζουμε ποιοι είναι οι υπάλληλοι που λαμβάνουν μπόνους και ποια είναι η κατανομή ανάμεσα στις διάφορες κατηγορίες των υπαλλήλων, διότι τα ποσά είναι πολύ σημαντικά. Διότι αν γνωρίζει κανείς ότι ε, κερδίζει κανείς ε, πάνω από 10.000 ε, ευρώ τον χρόνο, το μπόνους μπορεί να ανέρχεται στα 40.000 ευρώ τον χρόνο. Λοιπόν, λοιπόν, το ποσό πολύ υψηλό. Θα ήθελα να μάθω πώς θα αντιμετωπίσετε αυτό το πρόβλημα στο μέλλον. Θα μπορούσατε, μάλλον θα κάνετε μια δημοσίευση όλων αυτών των στοιχείων είναι ένα ερώτημα το οποίο θέσαμε και το 2010 στο πλαίσιο της έκθεσης για την, αναβολή, για την απαλλαγή. Ε, κάτι ακόμα, για μια σειρά ερωτήσεων η τράπεζα μας παραπέμπει στο θέμα της, ε, των ε, απορρίτων ε, πληροφοριών θα έχουμε κάποια εξέλιξη το 2013, το 2014, το 2015. Και τελευταία ερώτηση, για ποιο λόγο η τράπεζα δεν εφάρμοσε την ε, ισότητα ανδρών γυναικών, ισότητα των φίλων. Λυπάμαι που ε, είναι πολλές οι ερωτήσεις που θέτω, ξέρω ότι έχετε λίγο χρόνο, αλλά τα θέματα είναι σημαντικά και πρέπει να ε, ληφθούν απαντήσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πριν δώσω το λόγο στους συζητητές, ε, θα ήθελα κυρία Μπάρτεν ε, να ε, τοποθετηθείτε εσείς και να σας ευχαριστήσω και για τις γραπτές ερωτήσεις που έχετε καταθέσει. Σας καλωσορίζουμε θερμά και έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε τη δυνατότητα να συμμετέχω στην απαλλαγή για το ε, Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης. Ε, υπάρχουν βέβαια ορισμένα πράγματα που αφορούν, πέρα, που αφορούν ε, πέρα από το ΕΤΑ και πέρα από τη δική μου αρμοδιότητα, οπότε μπορεί να μην είμαι η, η μεγαλύτερη αρμόδια για, την, για ορισμένες απαντήσεις για τα βόνους. Αυτό που θα ήθελα να κάνω, δεδομένου ότι δεν έχουμε και πολύ χρόνο πλέον, ε, αν θέλετε το 2011 σε μία από τις τακτικές επισκέψεις στο ελεκτικό συνέδριο να ε, έρθετε σε επαφή μαζί μας, να έχουμε λίγο χρόνο να σας συναντήσουμε και να απαντήσουμε σε ερωτήσεις κυρίως ε, για την εξωτερική δανειοδότηση. Μπορώ να δώσω λίγο περισσότερο χρόνο για μία κάπως πιο ανεπίσημη συζήτηση. Επίσης, ε, θα ήθελα να πω ότι είναι η πεντηκοστή επέτειος ε, της δανειοδότησή μας στις χώρες ΑΚΕ. Θα υπάρξουν κάποιοι εορτασμοί μαζί με τις ε, υπόλοιπες επιτροπές αρμόδιες θα προσκληθείτε κι εσείς. Για ορισμένα ζητήματα τώρα που θέσατε ερωτήματα, με ρωτήσατε ποια είναι η άποψή μας για το κατά πόσο αυτό θα πρέπει να αποτελέσει τμήμα της επίσημης χορήγησης απαλλαγής. Δεν χρειάζεται. Ε, θέλουμε να λογοδοτούμε βέβαια και να είμαστε υπόλογοι. Ο μόνος λόγος που δεν συμμετέχουμε σε αυτή τη διαδικασία είναι γιατί το ΕΤΑ δεν είναι τμήμα του προϋπολογισμού, εκτός αν δεν κατάλαβα καλά την ερώτησή σας. Θα θα είχαμε ένα πρακτικό πρόβλημα με τη συμμετοχή του ΕΤΑ στον προπολογισμό για τον, για, λόγω του τρόπου με τον οποίο δουλεύει με την διευκόλυνση την επενδυτική. Αν ε, ήμασταν τμήμα του προπολογισμού το 2020 μέχρι το 2020 θα χρειαζόμασταν κάποιο είδους χρηματοδότηση για να μπορέσουμε να διατηρήσουμε και εμείς τη χρηματοδότησή μας στις άλλες χώρες. Ε, ε όσον αφορά το ερώτημα τώρα περί διαφάνειας, ε, Είμαστε στη μέση των ε, ε, της ανάπτυξης ε, μηχανισμός, ε, γιατί, μηχανισμό, γιατί οι περισσότεροι φορείς που συμμετέχουν είναι λιγότερο διαφανείς λόγω απορρίτων τραπεζών, όπως είπα. Πιστεύω όμως ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε καλύτερα και θα ήθελα πάρα πολύ του χρόνου να ξανάρθω να σας παρουσιάσω μια βελτίωση στην κατάστασή μας, παρά το γεγονός ότι προσπαθούμε πάρα πολύ να επιτύχουμε τα επίπεδα της Παγκόσμιας Τράπεζας. Η Ευρωπα ευρωπαϊκά όργανα μερικέ φορές μειώνουν τη διαφάνεια εντός οποία λειτουργούμε και αναφέρομαι κυρίως στον επόπτη προστασίας ε, ε, δεδομένων. Ίσως θα μπορούσαμε να συμμετέχουμε στη Διεθνή Πρωτοβουλία Περί Διαφάνειας, αν προσχωρήσουμε στη συγκεκριμένη προσπάθεια, ε, όμως για την ώρα δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό γιατί τα πρότυπα αφορά, αφορούν κυρίως ε, ε, ε φορείς ε, που δίνουν επιδοτήσεις. μπορώ να σας πω περισσότερα ίσως του χρόνου όταν θα έχουν εξελιχθεί τα πράγματα. Αυτά σε σχέση με τη διαφάνεια. Με μπέρδεψε λίγο η ερώτηση για το ποιε χώρε Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσαν να δημιουργήσουν προβλήματα όσον αφορά τη φορολογία. Κοιτάξτε, εμεί δεν μπορούμε απλώς ε, να κρίνουμε από μόνοι μας ποια δικαιοδοσία είναι φορολογικός παράδεισος. Πρέπει να δούμε ποιος, ε, ε, να δούμε τι γίνεται στον όσα, να δούμε τέλος πάντων τι μη συνεργάσιμες δικαιοδοσίες, ε, γιατί υπάρχουν κάποιες που είναι αδύναμες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και είναι αναπτυσσόμενες χώρες ε, και, σε, από οικονομικής και από κυβερνητικής απόψεως. Επί της αρχής λοιπόν πρέπει να πούμε ότι ναι, δημιουργούνται κάποια προβλήματα, έχουμε πολύ λιγότερο αυστηρές προδιαγραφές για εκείνους από ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά τις ρήτρε για τις συμβάσεις και τον περιορισμό ορισμένων προβλημάτων αλλά μπορεί να μην κατάλαβα καλά την ερώτηση και αν θέλετε να σας ξαναπαντήσω αν δεν κατάλαβα καλά. Όσον αφορά τώρα σε ε, περιπτώσεις ε, ε, διαφθοράς, σε όλες τους οργανισμούς ε, που έχουν βελτιωθεί στα συστήματα και έχουν εισαγάγει πάρα πολύ, που έχουν εισαχθεί πολύ, έχει, πολύ, έχει εισαχθεί πολύ ευαισθητοποίηση και κατάρτιση σχέση με αυτό το θέμα. Ε, διαπιστώνονται τέτοιε περιπτώσεις, όχι επειδή υπάρχει περισσότερη διαφορά από ό,τι στο παρελθόν, αλλά γιατί η μέθοδος ανείχνευσής τους είναι καλύτερη. Οπότε νομίζω ότι καταρχήν αυτό είναι κάτι καλό. Είναι ένα καλό σημάδι, δεν είναι κακό σημάδι αυτό, όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα τώρα είναι κάτι στο οποίο έχω δει να σημειώνεται πρόοδος από τότε που ανέλαβα καθήκοντα και χαίρομαι όλος ιδιαίτερος που είδα τέτοιου είδους βελτίωση. Είχαμε μία επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα της Αμνηστίας και ήταν και άλλοι επιρρογνώμονες από άλλους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς να μας πούνε ακριβώς τι κάνουν σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα και με καθησύχασε κάπως το γεγονός ότι πιστεύαμε ότι καθυστερούσαμε αλλά χάρη σε πίεση από ανθρώπους σαν και όχι δεν έχουμε καθυστερήσει και τόσο πολύ για τα ανθρώπινα δικαιώματα γιατί έχουμε μια τέτοιου είδους προσέγγιση ε, στι κατευθυντήρες γραμμές ε, κοινωνικής αξιολόγησης. Απλώ το θέμα είναι πώ θα το συνδέσουμε με τις ε, διάφορες κατηγορίες που είναι αντικείμενα των εκθέσεων. Υπήρξε πάντω ιδιαίτερη πρόοδο, πολύ μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση σε σχέση με το θέμα αυτό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μεταξύ του προσωπικού. Δεν είμαστε βέβαια τέλειοι ακόμη για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά τέλος πάντων ε, ε, το πλαίσιο μας βοηθά πολύ περισσότερο. Όσον αφορά τώρα τη δημοσίευση των πόνους, όπως είπα προηγουμένως, ε, δεν έχουμε πόνους, έχουμε βραβεία επιδόσεων. Ε, ε, έτσι επιβραβεύουμε την καλύτερη επίδοση. Δεν ξέρω κατά πόσο υπάρχουν κάποια σχέδια δημοσίευση αυτών των βραβείων, για να το πω έτσι. Εγώ δεν το γνωρίζω, οπότε δεν μπορώ να σας δώσω καλύτερη απάντηση αυτή τη στιγμή. Μπορώ να σας δώσω όμως μια λεπτομερέστερη γραπτή απάντηση, αν θέλετε. Όσον αφορά τώρα τα αποτελέσματα και πότε θα φανούν από εμά. Ελπίζω να, λάβατε, να πήρατε μία γεύση της έκθεσης της σχετικής που για πρώτη φορά ε, ε καταρτίζει σχέση με αυτό το θέμα δείχνει ότι χρειαζόμαστε πολύ χρόνο για σημαντικά αποτελέσματα για να φανούν σημαντικά αποτελέσματα. Χρειάζεται δηλαδή πολλής χρόνος, πολλά χρόνια για να δούμε μια σοβαρή μείωση της φτώχειας. Ε, προσπαθούμε με έμεσο τρόπο να επιτύχουμε τη μείωση της φτώχειας, όπως ας πούμε με την αύξηση της απασχόλησης και μπορεί να χρειαστούν πάρα πολλά χρόνια για να αρχίσει ας πούμε ένας μηχανισμός ιδεοδότησης να δουλεύει. Πολλές φορές μας ρωτούν επίσης για τον οικονομικό τομέα ειδικότερα και τη διαφάνεια και ε, τη διαφάνεια της ε, χρηματοδότησης των τελικών δικαιούχων. Έχουμε παραδείγματα τεσσάρων προγραμμάτων στη ΣΑΚΕ, σας πούνε καλύτερα τα παραδείγματα αυτά. Περισσότερα από όλα αυτά μπορώ να σας πω εγώ. Ελπίζω ότι να έχουμε και τις σχετικές εκθέσεις σύντομα διαθέσιμες. Έχουμε βέβαια και τη δική μας άποψη για το πώς μπορούν να βελτιωθούν τα πράγματα. τελευταία ερώτηση, πάλι δεν την κατάλαβα πολύ καλά. Τι εννοούσατε ακριβώς, μιλούσατε για το θέμα των ανθρωπίνων πόρων που δεν είναι δικής μου μιλήσατε γιατί ακριβώς, για την ισότητα, γιατί ακριβώς μιλήσατε. Ε, Κοιτάξτε, ε, ο συνάδελφος Μπέρμαν είναι στον κατάλογο. Αν μου επιτρέπετε θα δώσω το λόγο σε άλλους συναδέλφους. Πρώτα. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ για τις απαντήσεις σας στις ερωτήσεις είχα ετοιμάσει μια ερώτηση σχετικά με την διαφθορά. Νομίζω όμως ε, ότι έχει ήδη εξεταστεί για να λυθεί παρόμοια ζητήματα. Έχει θίξει ένα συνάδελφο γι' αυτό λοιπόν προκειμένου να ξεκονομήσουμε χρόνο δεν θα επιμείνω. Ευχαριστώ. Κύριε Μπέρμαν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Δεν έχουμε στην διάθεσή μας άλλο του Γερμανείς, επειδή και αυτοί θέλουν πολύ σωστά να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Για το θέμα τώρα της ε, Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, θα ήθελα να το αφήσω κατά μέρος ε, γιατί έχει εξεταστεί σε άλλα, σε άλλα βήματα. Τώρα το ζήτημα του ε, βιομηχανίας αλουμινίου στη Μοζαβίκη που συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και άλλους να πω ότι πρόκειται και για ένα άλλο πρόβλημα το οποίο προέκυψε και αφορά την εξαγωγή συναλλάγματος από την Μοζαβίκη θα μπορούσαν να πούν ότι η Μοζαβίκη είναι μέτοχος, ναι, αλλά δεν ε, εισπράττει αυτά τα οποία θα έπρεπε να εισπράττει ως ε, μέτοχος της ε, επιχείρησης. Η ΕΤΕ έχει σκεφτεί το ζήτημα το, το ζήτημα της ισότιμης ανάπτυξης θα πρέπει να βασίζεται ε, στις αποφάσεις που λαμβάνει η τράπεζα προκειμένου να συμμετάσχει σε κάποια προγράμματα ή όχι. Ο κ. Μούλντερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Η ερώτησή μου είναι παρόμοια με την προηγούμενη για το νέο χρηματοδοτικό μέσο. Ας υποθέσουμε ότι η ΕΤΕ παρέχει εγγύηση σε κάποια χώρα προκειμένου να μπορέσει να αναπτύξει την οικονομία της. Πώς ε, λειτουργεί αυτή η εγγύηση. Πώς η τράπεζα μπορεί να εγγυηθεί ότι τα κονδύλια δεν θα πάρουν έναν διαφορετικό δρόμο από τον αρχικό, από τον, αυτό που είχε προβλεφθεί. Επειδή όμως πρόκειται για τραπεζική εγγύηση, θα είναι εύκολο να υπάρξει κάποια εκτροπή τουλάχιστον ενό τμήματο. Ευχαριστώ. Και σα δίνω το λόγο, κυρία Μάρτιν. Ε, κοιτάξτε, να τα πω γρήγορα, αλλά κάτι να πω τουλάχιστον από το τίποτα καλύτερο και από το. Κοιτάξτε, ε, όσον αφορά την ε, επιλεξιμότητα, θέλω να πω ότι όταν ε, χρηματοδοτήσαμε αυτό το project στη Μοζαμβίκη, τότε δεν ήμασταν τόσο αυστηροί όσο είμαστε τώρα. Και ένας από τους δείκτες ε, σε αυτό το πρόγραμμα έχει σχέση με τα δημοσιονομικά έσοδα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να ε, συμπληρώσει κανείς αυτό το στοιχείο. Εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε. Βεβαίως οι εξορίξεις είναι ένας με πάρα πολλές διακυμάνσεις, αλλάζουν οι τιμές ε, των πρώτων υλών. Εν πάση περιπτώσει, ε, ε, σε τελική ανάλυση δεν έχουμε χρηματοδοτήσει τέτοιου είδου project από το 2007. Αυτή είναι η απάντησή μου. Όσον αφορά το νέο χρηματοδοτικό μέσο, εγώ δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία μεγάλη πρόκληση όσον αφορά τις εγγύσεις, γιατί σε τελική ανάλυση όλα έχουν την τιμή τους και για εμά και για την αγορά. Και ακόμα και αν υπάρχει κάποια εγγύηση και αυτή κοστίζει. Δεν θα έλεγα λοιπόν ότι εδώ δεν είναι απαραίτητο να γίνεται λεπτομερής ε, έκθεση και να μην ισχύουν οι κανόνες περιγγύσεων. Ισχύουν τα ίδια. Πρόεδρος, ξέρω ότι δεν έχουμε αρκετό χρόνο για να μπούμε σε λεπτομέρειες ε, και γι' αυτόν τον λόγο δώσαμε και τη δυνατότητα να δοθούν ε, γραπτές ε, ερωτήσεις. Δεν μπορούσαμε να αποφύγουμε τη συζήτηση με τον Επίτροπο κύριο Σέμετα. Ευχαριστώ την κυρία Μπάρτον και όλη του ομάδα του συνεργάτες της που ήρθατε εδώ, που απαντήσατε στις ερωτήσεις μας και θέλω να υπενθυμίσω σε όλους σας ότι υπάρχει μια πρόσκληση εμείς, η Επιτροπή μας, έχουμε καλέσει όλους ε, για μια άτυπη έτσι συνάντηση και εκεί μπορούμε να τα πούμε. Και ε, τέλος θα κλείσει τη συνεδρίση ο εκπρόσωπος του ελεγκτικού συνεδρίου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, θα είμαι πάρα πολύ σύντομος. Χαίρομαι πάρα πολύ που θα σας παρουσιάσω έκθεση. Ε, το συνέδριο έχει εξετάσει τις ε, διάφορες συστάσεις και λόγω του ότι βέβαια δεν υπάρχει, μάλλον έχει περάσει πολλή χρόνο από τότε που δημοσιεύτηκαν οι εκθέσεις, η έκθεση καλύπτει τρεις τομείς ε, και συνολικά 51 συστάσεις, εκ των οποίων οι 45 εξακολουθούν να θεωρούνται σημαντικές. Θέλω λοιπόν να σας επισημάνω ότι το ε, ελεγκτικό συνέδριο ακολουθεί τις δικές του συστάσεις ε, και όχι αυτές ε, του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και θα ήθελα να ξέρω κατά πόσον συμφωνείτε ή μήπως πιστεύετε ότι στην έκθεση που θα συντάσσουμε κάθε χρόνο κατά πόσον εκεί θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας και τα αιτήματα του ε, Κοινοβουλίου. Ε, βεβαίως δεν θέλω να σας αντιμετωπίζουν διαφορετικά. Συνέβη αυτό και σκεφτήκαμε ότι θα πρέπει να δούμε καταρχήν ε, τις ε, δικές μας τις ε, συστάσεις. Γι' αυτό λοιπόν, όπως ε, σας είπα, με μεγάλη χαρά, όταν θα έχετε ολοκληρώσει την έκθεσή σας, να μας πείτε ε, σε μένα που είμαι εισηγητής, τι, πώς ακριβώς θα πρέπει να, το, να εξελιχθούμε σε αυτό το θέμα. Δεν νομίζω ότι έχω να προσθέσω τίποτα άλλο. Έχετε δει τα στοιχεία και όπως σας είπα, αυτή η ετήσια έκθεση θα γίνεται κάθε χρόνο, γιατί δεν αρκεί μία έκθεση ελέγχου. Πρέπει και μετά να δούμε τι ακριβώς έκανε η Κομισιόν, αν ακολούθησε τη συστάση μας. Κάθε χρόνο λοιπόν θα ερχόμαστε εδώ και θα παρουσιάζουμε μία ε, έκθεση με βάση τα πεπραγμένα. Πρόεδρος. Συγητής, θέλετε το λόγο. Έχει περάσει πολλή ώρα. Θα σημειώσω την πρόταση του ελεγκτικού συνεδρίου. Νομίζω ότι είναι ενδιαφέρουσα πρόταση. Θα ήταν χρήσιμο να συμπεριληφθούν οι συστάσεις ε, της ε, Επιτροπής μας ε, όταν θα αξιολογήσουμε τι συνέβη τα τελευταία χρόνια. Δεν μπορώ να μιλήσω εκ μέρους βέβαια όλη της Επιτροπής. Πρέπει να περιμένουμε τη συνεδρίαση των συντονιστών, αλλά μου φαίνεται μια καλή πρόταση. Μπορούμε να τη λάβουμε υπόψη για το μέλλον. Τα υπόλοιπα θα πρέπει να τα υποβάλουμε γραπτός. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Τράπεζα Επενδύσεων που ήρθε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ στους, τους συναδέλφους που επέδειξαν πειθαρχία. Ευχαριστούμε το Ελεγκτικό Συνέδριο και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Ευχαριστούμε τη Γραμματεία και τους μεταφραστές και τους διερμηνείς που τους καθυστερήσαμε. Λοιπόν, στην πέμπτη, στον πέμπτο όροφο θα γίνει η δεξίωση. Αν θέλετε να έρθετε, ε, θα χαιρόμουν πολύ να μπορώ να έχω την δυνατότητα να σας ε, υποδεχθώ στον πέμπτο όροφο. Γεια σας.